So, Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, επαναλάβουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε τρεις ψηφοφορίες σήμερα. Το ένα είναι η τροποποίηση των οδηγιών όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να αντεθούν στην Επιτροπή. Μετά έχουμε το backloading το λεγόμενο και μετά μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Βιομηχανίας για ενέργεια πανενεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας. Και μετά έχουμε τη συζήτηση λεπτομέρειες επίτευξης του στόχου του 2020 για τις μειώσεις εκπομπών από καινούργια γεωταχή. Και το απόγευμα έχουμε τις ακροάσεις διάφορα θέματα, το σημείο 10, τύχη βορειοανατολικός Ατλαντικός ε, και τελευταίο σημείο το απόγευμα είναι η διάθεση στην αγορά φορητών μπαταριών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για σύρματα ηλεκτρικά εργαλεία. Και έχουμε την ακρόαση του Hans Breinix, νέου εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Και παρακαλώ τους να είναι παρόντες για να ξεκινήσουμε στις 3 η ώρα με γεμάτη αίθουσα όπως τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με την οδηγία του πρωινού και εδώ πέρα έχω εγώ την τιμή να είμαι εισηγητής. Ξεκινάμε με το άρθρο 1, τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Όχι, έχει καταπέσει αυτή που λέτε. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κυρία Κονή. Έχω ένα πρόβλημα, με... πρόβλημα μετάφρασης. Έχουν μπερδευτεί τα νούμερα 15, 16, 6, 5, τα κανάλια της Διερμηνίας έχουν μπερδευτεί, λέει η κυρία. Η 4 έγινε δεκτή και άρα οι 15 και οι 16 έχουν καταπέσει. Ψηφίσαμε την 5, επίσης έχει δεκτή και πέρασαμε στην 6 την οποία επίσης ψηφίσαμε, επίσης έγινε δεκτή και μετά συνεχίζουμε με την υπαριθμόν 7. Εντάξει. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε λοιπόν στην ε, ενοποιημένη 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 και 22 αυτός είμαι σπέρ κατά αποχές δεκτές 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά. Για την πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 64 υπέρ. Περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος και πάλι ηλεκτρική. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Και θα ζητήσω και μία έντολη. Σας ευχαριστώ. Έντολη λοιπόν για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ε, σύντομα τη συζήτηση με το Συμβουλίο και αυτή η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, αρχή τη ψηφοφορία. Πέρας. 62 υπέρ μια αποχή. Σας ευχαριστώ για την ε, εμπιστοσύνη σας. Ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με το Συμβούλιο και μάλλον θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Οπότε Για την επόμενη ψηφοφορία. Θέλω να ζητήσω ονομαστική ψηφοφορία για τρία σημεία. Το ένα είναι η απόρριψη της πρότασης, τροπολογία 11 που αλλάζει νομική βάση και την τελική ψηφοφορία. Θέλω να ζητήσω για αυτά τα τρία σημεία ονομαστική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πρώτον, δηλαδή, για το πρώτο μπλοκ για την απόρριψη, μετά για τροπολογία 11, για την νομική βάση δηλαδή, και τις δύο, και τις δύο τελικές ψηφοφορίες. Ακριβώς, λέει ο κύριος Άικχαουτ. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του, να σηκωθεί, με συγχωρείτε. Εντάξει, αρκεί 30 υπέρ. Οπότε 18 θα ήταν ο απαιτούμενος αριθμός. Οπότε το πρώτο μπλοκ, η τροπολογία 11 και οι δύο τελικές ψηφοφορίες θα γίνουν ηλεκτρονικά. Έχουν όλες τις κάρτες ε, για την ψηφοφορία. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως με το πρώτο μπλοκ προτείνω να ψήσουμε ηλεκτρονικά γιατί μόλις το συμφωνήσαμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 υπέρ, 40 κατά, 2 αποχές. Δεν γίνεται δεκτό το πρώτο μπλοκ. δεν χρειάζονται χειροκροτήματα ούτε και από τους ε, προσκεκλημένους και θεατές. Ερχόμαστε στην τροπολογία 30, Βίλτς, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32, υπέρ, Κατά. εποχές Απορρίπτεται. Συμβε... Ενοποιημένη 1. Συγγνώμη. Ηλεκτρονικά. Ενοποιημένη ένα Ώστε να μην υπάρξουν ε, αμφισβητήσεις. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Το ΕΛΚ έχει ένα που ψηφίζει παραπάνω. Ξεκινάμε και πάλι. Πάλι από την αρχή. Ενοποιημένη τροπολογία 1. Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. Πάλι υπάρχει ένας παραπάνω που ψηφίσει από, την, τάξει του ΕΛΚ. Και πάλι πρέπει να ξεκινήσουμε. Για τρίτη φορά ξεκινάμε για την ενοποιημένη 1 ε, ηλεκτρονικά μέσα. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας. 49 υπέρ 16 κατά γίνεται δεκτή η τροπολογία. Τροπολογία 39 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 40 με 26 γίνεται δεκτή σαφώς. 11. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27 υπέρ 38 κατά απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένοι 2. Ηλεκτρονικά προτείνω άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 47-19 γίνεται δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία 5. <clears throat> Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές Δεν είναι σαφές. Κάνουμε έλεγχο για την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 28 υπέρ 38 κατά απορρίπτεται 27 <clears throat> υπέρ κατά αποχές και εδώ δεν είναι σαφές κάνουμε έλεγχο σφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 27-38 28 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές και εδώ δεν είναι σαφές έλεγχος για την 26 ψηφίσατε όλοι πέρας 45 υπέρ 21 ψήφι κατά γίνεται δεκτή σαφώς η πρώτη ψηφοφορία με ονομαστική κλίση το σύνολο του, της έκθεσης, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 38 υπέρ 26 κατά μία αποχή γίνεται δεκτό το σχέδιο έκθεσης και θα καταγραφεί φυσικά και η ονομαστική ψηφοφορία. Η δεύτερη ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πάλι 38 υπέρ 25 κατά με δύο αποχές. Γίνεται λοιπόν <clears throat> δεκτή και θα ήθελα να σας ζητήσω μια σύντομη διακοπή για να μπορέσω να συνεννοηθώ με τους συντονιστές ένα λεπτό και μετά θα περάσουμε στη συνέχεια.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 So, ich bitte alle wieder Παρακαλώ ξανακαθίστε. Και η νέα διαδικασία για την έγκριση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο αποφασίσαμε με τους ε, συντονιστές να καταλήξαμε στο ότι πρέπει να κάνουμε μία ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν μία ανάγκη να έχουμε μία σαφή εικόνα για τη θέση της Επιτροπής μας, γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας για το αν θα πρέπει να έχουμε ε, εντολή διαπραγματευτική. Χρειάζονται 35 συνάδελφοι να υπερψηφίσουν. Αν δεν υπάρξει συμφωνία θα πρέπει να πάμε στην Ολομέλεια. Και υπάρχουν ορισμένοι που θέλουν να λάβουν το λόγο τώρα σχετικά. Ο Πέτερ Λίζε πρώτα. Μία παράκληση να το ξανασκεφτούμε. Ξέρω ότι πολλοί θεωρούν ότι εμείς είμαστε η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για τα θέματα αυτά δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα η Επιτροπή Ήτρε για τα θέματα των, το, της κλιματικής αλλαγής. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτούς οι οποίοι λένε ότι πρέπει εμείς να αναλάβουμε την ευθύνη για αυτά τα θέματα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι αν μας βοηθάει στο μέλλον να οικοδομήσουμε μια λογική πολιτική για την ενέργεια και τα κλιματικά. Δεν το ξέρω αυτό. Ε, γι' αυτό σας ζητώ να το ξανασκεφτούμε και ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα να καταλήξουμε σε μια πρόταση και την επόμενη εβδομάδα έχουμε συνεδρία τη Επιτροπής, μπορούμε να επανέλθουμε εκεί και να ψηφίσουμε, γιατί το θέμα αυτό είναι ήδη πολιτικά αμφιλεγόμενο και ίσως θα πρέπει να συνεννοηθούμε και με τους συναδέλφους με την Επιτροπή Ήτρε για να δούμε κατά πόσο είναι διαθέσιμοι να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Αν δεν θέλουν, τότε πάλι θα είναι το τελικό αποτέλεσμα το ίδιο. Αλλά αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση, ίσως θα είναι επωφελέστερο για όλους. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω αυτούς που ζήτησαν, που έχουν καταθέσει αυτή την τροπολογία, να μην κάνουν τώρα την ε, ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι επίμαχο το θέμα και πάρα πολύ σημαντικό για πολλές χώρες και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το ψηφίσουμε, να ψηφίσουν όλα τα μέλη και έτσι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να δώσει εντολή για διαπραγματεύσεις. Δεν θα πρέπει να έχουμε μια ε, μικρή ομάδα να αποφασίσει. Είναι σημαντικό για τη βιομηχανία, για το μέλλον της Ευρώπης και δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Ο κύριος Ντέιβις. Η ομάδα μου δεν είχε δυνατότητα να το συζητήσει, δεν ήταν στον κατάλογο ψηφοφορία. Αν είναι δικαστικά δυνατό να καθυστερήσουμε, δεν έχω πρόβλημα να ακολουθήσουμε το τελίζα την πρόταση. Μια εβδομάδα δεν κάνει διαφορά, θα πάμε και πάλι στην Ολομέλεια. Εάν θέλουμε να υποστηρίξουμε παραπομπή στην ε, Ολομέλεια. Απ' την άλλη πλευρά, είναι κρίσιμο θέμα αρχή. Κατά πόσο το θέμα πρέπει να πάει στην Ολομέλεια και να ψηφίσει όλο το Κοινοβούλιο πριν στι διαπραγματεύσει. Απ' την άλλη, αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Όλο το μέλλον της προσέγγισης στην αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από αυτό και το Συμβούλιο ήταν διερημένο. Θα ήταν καλό αν θα μπορούσαμε να βρούμε ε, κάποια συμφωνία με το Συμβούλιο όσον αφορά τη μελλοντική προσέγγιση και να το ψηφίσουμε αυτό στην Ολομέλεια. Πρέπει να βρούμε την ε, ισορροπία που είναι πολύ λεπτή και χρειαζόμαστε ή δυνατόν περισσότερο χρόνο για συζήτηση. Uh, είναι προφανέστατο ότι το κοινοβούλιο στο σύνολό του είναι διχασμένο οπότε δεν είναι σωστό να διαπραγματευόμαστε όταν uh, δεν έχουμε ένα σαφές μήνυμα από την uh, Ολομέλεια. Είχαμε και άλλες ε, τέτοιες δύσκολες καταστάσεις όπως ε, στο Ρίτς. Τα υπόλοιπα είναι σαφή. Έχει η Επιτροπή μας δικαίωμα να πάει στη διαπραγμάτευση, αλλά τελικά, και θεωρώ πως είμαι αρκετά ουδέτερος, πρέπει να ξέρουμε πως θα έχουμε και εδώ μέσα πλειοψηφία για να πάμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Οπότε έχει δίκιο ο Πετρελίζε. Ας το ξανασκεφτούμε και ίσως μπορέσουμε να βρούμε κάποια αριθμίση για να έχουμε ευρύτερη διαπραγματευτική βάση. Οπότε εγώ θα πρότεινα να ε, περιμένουμε μία εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει. Μήπως βρεθεί κάποιο συμβασμός. Νομίζω πως τέλος θα είναι καλύτερα. Μάλιστα. Νομίζω πως είναι σαφές. Δεν θα ε, ψηφίσουμε σήμερα. Θα το ξαναδούμε με τους ε, σκιώδεις συγητές και δεν ανάγκη να πάμε με μία ψήφο διαφορά Οπότε η ψηφοφορία αυτή ολοκληρώθηκε και πάμε παρακάτω στο κείμενο. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Συνεχίζουμε με το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Που αφορά τη γνωμοδότηση για την Ήτρε και πρέπει να σας πω πως είναι η γνωμοδότηση της κυρίας Κούκοβιτς και η τροπολογία 33 του κυρίου Περελαιό Ροντρίγκες αποσύρθηκε. Να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 3 υπέρ οι κύριοι και οι κυρίες ε, οι λομπίστες εκεί πέρα στο βάθος που ε, έχουν άλλη μία εβδομάδα χρόνο για να κινητοποιηθούν θα μπορούσαν ίσως να κάνουν λίγο ισχύα σας Παρακαλώ λοιπόν να μεταφερθούν έξω οι συζητήσεις για να ψηφίσουμε την έκθεση Κουκουβίτ. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5-2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Το δεύτερο μέρος της 5. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 31, 31 υπέρ, 30 κατά. Δεκτή. 7 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 8-1 Αναρός Μπαχτέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 να επαληθεύσουμε την 13 αρχιετή ψηφοφορία Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Θα την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 31, 32 απορρίπτεται. 15 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην 16 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Θα το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 19 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18-1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18 μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές, θα το επαληθεύσουμε. Τη 23 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ξεκάθαρα γίνεται δεκτή. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και περνάμε στην 22 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ να επαληθεύσουμε την 25 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή σαφώς 26 υπέρ κατά εποχές δεκτή να την επαληθεύσουμε δεν είμαι σίγουρος κι εγώ ψήφισαν όλοι πέρας ε, πρέπει να ξαναψηφίσουμε ξανά την 26 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Mm Πέρας. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Φαίνεται πως έχει γίνει δεκτή. Ε, 36 υπέρ. Υπέρ της 36 κατά εποχές δεκτή να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή λοιπόν. 38 τώρα υπέρ. Κατά. Έξι συνάδελφοι ε, ψήφισαν. 38 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Επαληθεύουμε την 40 θέλει η συγγήτρια. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Θα την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απόρριπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. 45 υπέρ. Το πρώτο μέρος. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Δεκτό. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Να επαληθεύσουμε την 47 αρχιετή ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. σοσιαλδημοκράτες. Κάποιος είναι παραπάνω. Λοιπόν, τώρα είναι εντάξει. Α, απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. 46 λοιπόν ηλεκτρονικά. Θα τα απολυθεύσουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. δεκτή. 48 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ναι, ναι. ευχαριστώ να την επαληθέψουμε. Ψήφισαν όλοι. Ξανά πρέπει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της 48 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 51 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 53 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 54 και 55 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 56 μέρος δεύτερο να, να υπαλληθεύσουμε την 56 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή 46 με 18 56 μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 μέρος τρίτο υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 63 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 64 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 65 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 66 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται και μετά περνάμε σε προφορική τροπολογία της κυρίας Ούλουσκοκ, Χάουκ, το έχετε και στον κατάλογό σας. Δεν το έχετε στον κατάλογό σας. Θα το διαβάσω. Ζητά από την αρχή του προϋπολογισμού αντί για κομισιόν. Όποιος ε, εμπιστεύεται λοιπόν την κυρία Χάου και συμφωνεί, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συνεχίζουμε με την 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή να επαληθεύσουμε την 69 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται σαφώς 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ. Κατά. Αποχές με την ίδια πλουσία απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης. άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 64 ε, υπέρ, μία κατά μία αποχή, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. 18 Μαρτίου ψηφοφορία στην Ήτρα και πιθανώς στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τις ε, ψηφοφορίες και... Und ich übergebe an... Και δίνω ε, την Προεδρία στον ε, συνάλφο τον κύριο Γκερμπράντι. Okay, Σας παρακαλώ, εσάς όσοι δεν θέλετε να συνεχίσετε την παραμονή στη συνεδρίαση, να κάνετε ησυχία ή αν θέλετε φύγετε από την αίθουσα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας, με την ημερήσια διάταξη. Θα συζητήσουμε την έκθεση του κ. Ούλμερ, λεπτομέρειε τη επίτευξη του στόχου μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα το 2020. Και θα ήθελα να δώσω στον κ. Ούλμερ το λόγο. Λίγη ησυχία σα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να αναφέρω τον στόχο αυτής της ε, πρότασης, όπως μπορείτε να κατανοήσετε. Από τον τίτλο και τις τροπολογίες, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος στα επιβατικά αυτοκίνητα με νέες μορφές ε, αυτοκίνησης που να είναι και οικονομικά και οικολογικά βιώσιμες. θα έχουμε ένα όριο από το 2015 130 ε, γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο και από το 2000 γραμμάρια το χιλιόμετρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους ε, στόχους και να συνεχίσουμε τη μείωση που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ε, ο στόχος μας είναι να υπάρξει μια μείωση 27% ώστε να μειωθεί η εκπομπή από τα μικρά αυτοκίνητα, αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει οι κατασκευαστές να αντιμετωπίσουν την ανάγκη εξέλιξη αυτοκινητών τα οποία θα είναι πιο πολυδάπανα στην σχεδίαση και την κατασκευή τους. Φυσικά οι νέες τεχνολογικές αλλαγές γίνονται κυρίως στα πιο μεγάλα αυτοκίνητα. Πρέπει να δοθούν όμως τα απαραίτητα κριτήρια και κίνητρα ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν περισσότερο νέες ε, ε, κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τα μικρότερα αυτοκίνητα. Ο στόχος μας είναι επίσης να εξασφαλίσουμε και μια δίκαια μορφή ανταγωνισμού μεταξύ των ε, αυτοκίνητων βιομηχανιών. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα το οποίο θα οδηγήσει σε καθυστέρηση της αγοράς νέων αυτοκινήτων. Η Κομισιόν επομένω πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν τη δυνατότητα να δουν αν μπορούν με εύκαμπτο τρόπο να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. και μέσα στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα πρέπει να καλύψουμε τα 15% της ε, μείωσης. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να καταλήξουμε στην επίτευξη ενός ε, στόχου 50 γραμμαρίων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε οι, κατα... οι καταναλωτές να επωφεληθούν από την επένδυση των αυτοκινητοβιομηχανιών σε εναλλακτικές μορφές κίνησης για τα αυτοκίνητα. Το καθεστώς αυτό κινήτρων θα εκπνεύσει το 2023. Θα είναι επίση απαραίτητο να υπάρξει μια τυποποιημένη διαδικασία δοκιμασίας ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα διαφορετικών ε, μοντέλων. Έχουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία η οποία θα πρέπει να αποτελεί μια ρεαλιστική <clears throat> απεικόνηση της ε, χρήσης των αυτοκινήτων και επομένως να κάνει μια σωστή επιλογή. Ζητούμε επίση από τους ε, αυτοκίνητο βιομηχανούς να επιτύχουν, να δημιουργήσουν μια βάση επί της οποίας μπορούν να εξασφαλίσουν την μείωση των εκπομπών ε, διοξιδίων του άνθρακος. Θα πρέπει να παρακινήσουμε και τις βιομηχανίες και τους ε, ε, υπεργολάβους και προμηθευτές τους να κάνουν όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να μειωθεί η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος και η κατανάλωση καυσίμου φυσικά ώστε με τον τρόπο αυτό να μειωθεί η συνολική επιβάλληση του περιβάλλοντος. Η διαδικασία πιστοποίησης προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχει προχωρήσει επαρκώς ώστε να παρακινήσει τη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογικών αντιλήψεων Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει, έχει σταθεί πολύ περιορισμένη η καινοτομία σε ό,τι αφορά την επίτευξη στόχων του περιβάλλοντος. <clears throat> Ένα παράδειγμα το οποίο μπορώ να σας δώσω είναι η χρήση ευφυών συστημάτων πλοήγησης που μπορούν <clears throat> να συνδυαστούν με υβριδικά αυτοκίνητα ώστε όταν να μπορεί να φορτιστεί η μπαταρία όταν αυτό είναι εποφελές από άποψη κατανάλωσης και αυτό θα οδηγήσει σε ένα κύκλο κατανάλωσης ο οποίος θα είναι πολύ πιο οικονομικός. Για την ε, υιοθέτηση τώρα των ε, νέων αυτών υποδειγμάτων αυτοκίνησης από τους καταναλωτές αυτό νομίζω ότι θα είχε νόημα να μην αποφασιστούν αυτά τα νέα μοντέλα ήδη, οι νέοι τρόποι αυτοκίνηση ήδη από το 2014, αλλά να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προοπτικές για την μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος και να μην καταλήξουμε να έχουμε ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα μεν τα οποία να τροφοδοτούνται από θερμικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας που και αυτοί ε, επιβαρύνουν το περιβάλλον. Και θέλω να σας ευχαριστήσω εξ αρχής για τις προτάσεις τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Ε, προσβλέπω στη συζήτηση με εσάς και ιδίως με τους κοιόδης Thank ευχαριστώ πολύ κύριε Ούλμερ. Θα κάνουμε ένα γύρο με τους κοιόδης εισηγητές, με τον κύριο Περίλο που το S&D ξεκινάμε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εν πρώτης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, ρήτημο κύριο Ούλμερ για την έκθεσή του και για τη δαθεσιμότητά του ε, να συνεργαστεί και για να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα της εκθέσεως. Αυτός ο κανονισμός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος ε, διότι αφορά ένα τομέα στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή απασχόληση που υπόκειται μεγάλη συστολή και ύφεση κυρίως στην εσωτερική αγορά. Να σκεφτεί τον τελευταίο χρόνο η πτώση ε, εγγραφής νέων ε, οχημάτων, καταγραφής νέων οχημάτων ήταν περίπου ένα εκατομμύριο μονάδες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση οχήματα 21ου αιώνα, για να έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη που θα είναι ανταγωνιστική, ε, πρέπει να δώσουμε κίνητρα για την παραγωγή και την εμπορευματοποίηση οχημάτων που είναι άκρος τεχνολογικά με χαμηλή κατανάλωση καυσίμων και με χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. Από τη μία πλευρά αυτό θα μπορούσε να είναι μοχλός ανταγωνιστικός Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τη ζήτηση για αυτού του είδους ε, τα οχήματα ε, που σε αυτή την φάση βλέποντας το κόστος ε, βλέπουμε ότι η ζήτηση είναι πολύ χαμηλή. Για να πετύχουμε λοιπόν τους στόχους για την α, μείωση του, την ακομπότητα του δεξιού του μέχρι το 2050 και ο τομέας των μεταφορών είναι το 20% των εκπομπών και πρέπει και ο τομέας αυτός να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών. Ο στόχος των 90 ε, μικρογραμμαρίων που είχε καθοριστεί για το 2009 ήταν ένας σωστός στόχος. Όχι μόνο γιατί θέτει στόχους μέχρι το 2050, αλλά ανοίγει και το δρόμο για μικρότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Και γι' αυτό ο στόχος των 95 γραμμαρίων δεν θα πρέπει να ε, αποδυναμωθεί και θα πρέπει να δοθούν διάφορα κίνητρα για τους κατασκευαστές για να παράγουν οχήματα με χαμηλές εκπομπές. Αρκεί όμως αυτοί να μην αποδυναμώσουν τους στόχους της προτάσεως και να μην, έχουν, ε, να μην υπάρχουν κίνητρα υπό τον τύπο κυρώσεων για την παραγωγή συγκεκριμένων οχημάτων που θα χρησιμεύουν στην επιτευχθών των στόχων. Χρειάζεται ουδετερό τεχνολογική στην παραγωγή. Θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο που ακολουθούμε μέχρι τώρα, η μείωση των εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη την εφικτότητα των μέτρων προτείνονται, την τεχνολογική. Και πώς μπορεί να απορροφήσει η αγορά τα νέα οχήματα με την πολύ χαμηλή κομπή καυσαρίων. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον καταναλωτή μέσω αυτού του κανονισμού στον καταναλωτή θα πρέπει να δίνονται ε, πραγματικές πληροφορίες όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου τάνθρακος. Αναφέρομαι στον κύκλο των κειμένων για τις εκπομπές, ένα σύστημα που έχει επικριθεί γιατί είναι πάρα πολύ ευέλικτο. Και έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας επίσης υπάρχει όσον αφορά ε, την πραγματική ε, απεικόνηση των στιθικών οδήγησης. Μέχρι τώρα το σύστημα που χρησιμοποιείται μπορεί ίσως να υποτιμά τις πραγματικές εκπομπές διοξιδίου του ανθρακούς και την κατανάλωση καυσίμων και θα μπορούσε να ευνοεί τεχνολογίες οι οποίες δεν είναι βέλτιστες ε, βάσει αναλύσεως κόστος ωφέλους. Εκτιμώ τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο ενός νέου κύκλου δοκιμών ε, που ε, θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια, ένα ορισμό του μέχρι το 2004 και να εφαρμοστούν τα μέτρα μέχρι το 2017 όσο Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αξιολόγηση συνεπειών να δει πώς μπορεί να παρέμβει ε, για να εφαρμόσει μια νομοθεσία μεταβατική τροποποιώντας τον κανονισμό των ισχύοντα τώρα. Κατανοώ ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα ερμηνείας ε, των ε, στόχων που τέσσερα τις προηγούμενες δοκιμές. Ε, θα έπρεπε να υπάρχει πίνακα συσχετισμών που θα αντικατοπτρίζει τα σωστά επίπεδα μειώσεων. Αυτός ο νέος πίνακας δεν θα πρέπει να οδηγεί σε στρέβλωση όμως της, της αγοράς δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάποιους ε, κατασκευαστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Περίλιο. Ο κύριος Ντέιβις είναι επόμενος, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινάω με το να αποτίσω φόρο τιμής στον, ε, στην, στα επιτεύγματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Νομίζω ότι έχουν κάνει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Πράγματι με την δική τους αξιολόγηση ήδη ήταν σημαντική αυτή η πρόοδος γιατί το 2007-2008 μας είπαν ότι πολλά από αυτά τα οποία έγιναν στη συνέχεια ήταν ανέφικτα. Αλλά έχουμε καταλήξει σε μια θέση για το, τις μέσες εκπομπές 160 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρωπος ανά χιλιόμετρο. Αυτή ήταν μια μέτρηση που έγινε περίπου το 2007 και τώρα είμαστε περίπου στο 130 σήμερα. Αυτό είναι χρήσιμο βέβαια για να αντιμετωπίσουμε την ε, αύξηση θερμοκρασία του πλανήτη και δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί στον τομέα των μεταφορών. Είναι πολύ σημαντικό όμω και για του Ευρωπαίου πολίτε στην Ευρώπη και αλλού που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με χαμηλότερο κόστο από ό,τι στο παρελθόν και κατά μέσον όρο δεν χρειάζεται να καταβάλουμε μεγαλύτερο τίμημα για αυτά τα αυτοκίνητα. Τα μέτρα τα οποία ε, είχαμε εισάγει, εισαγάγει στο παρελθόν θα αύξαναν σημαντικά τις τιμές των αυτοκίνητων. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα τέτοιο και τα στοιχεία αυτά μπορεί να τα διακριβώσει και να τα επιβεβαιώσει και η Ένωση Αυτοκίνητων Βιομηχανιών στην Ευρώπη. Αυτό βέβαια οφείλεται στον ανταγωνισμό. Λεγόταν ότι υπήρχε υπερβολική ε, παραγωγή στον τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία και η αγορά θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Ναι, υπήρξε πρόοδο, αλλά πρέπει να γίνει και περαιτέρω πρόοδο. Νομίζω το να θέσουμε να θεσπίσουμε μακροχρόνιου στόχου ήταν κάτι που βοήθησε τι αυτοκινητοβιομηχανίε να έχουν σαφεί κατευθύνσει προ τι οποίε θα πρέπει να κινηθεί η καινοτομία και η πρόοδο και μπόρεσαν οι ερευνητέ και οι μηχανικοί να μπορέσουν να ακολουθήσουν μια σαφή πορεία. Εμεί θέσαμε το στόχο των 95 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο για πρώτη φορά το 2007 όταν το Κοινοβούλιο είχε περάσει την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τα θέματα αυτά. Πάρα πολύ λίγοι ήταν αυτοί που διαφυσβήτησαν αυτό το στόχο ακόμα και από το βιομηχανικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα 95 γραμμάρια μέχρι το 2020 μπορούν να επιτευχθούν με συμβατικές τεχνολογίες αυτοκίνησης. Και οι κατασκευαστές ε, ε, συστατικών στοιχείων για τους κινητήρες και τα αυτοκίνητα που απασχολούν περισσότερο κόσμο από τους συναρμολογητές των ε, κινητήρων μας είπαν ότι και αυτοί θεωρούν ότι η στόχη αυτή είναι εφικτή και επιτεύξιμη. Μετά από μερικά χρόνια λοιπόν όμως πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος μακροχρόνιος στόχος και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θεσπίσουμε ένα στόχο για το 2025. Μπορεί να θέλουμε να βγούμε <clears throat> από τους στόχους που είναι απλώς και μόνο στόχοι εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος κάποια στιγμή. Νομίζω στη, προς το παρόν όμως ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους να επιτευχθεί πρόοδος. Γιατί δεν μονάχα μείωση της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος είναι πρώτα απ' όλα μια βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης καυσίμων από αυτοκίνητα και αυτό ενδιαφέρει το μέσο οδηγό περισσότερο απ' όλα. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα στόχο 70 γραμμαρίων το χιλιόμετρο για το 2025 είναι κάτι το εφικτό και αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα για το οποίο θα πρέπει να αγωνιστούμε εμείς με τη δυνατότητα μετά από 3-4 χρόνια να κάνουμε μια εκ νέου επισκόπηση για να δούμε και τις νέες τεχνολογίες πλοήσης. Για τα super credits εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ρόλο, θα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα στη βιομηχανία για να αναπτύξουν αυτοκίνητα με πολύ χαμηλή εκπομπή διοξίδιου του άνθρακος Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα με μορφή χορηγήσεων, με ρυθμιστικές ε, διατάξεις οι οποίες θα βοηθήσουν αυτή την πορεία. Υπάρχει λοιπόν ένα ρόλος για τα super credits, αλλά δεν πρέπει να έχουν τέτοιο χαρακτήρα ώστε να στρεβλώσουν τους στόχους για τις εκπομπές που έχουμε θεσπίσει. Και όπως λέει και ο κύριος Σούλμερ στην έκθεσή του και ξέρω ότι είναι ανοιχτό για διαπραγματεύσεις, ε, ίσως είναι υπερβολικό να βασιστούμε μόνο σε αυτά τα super credits. Για τον κύκλο δοκιμασιών τώρα. <clears throat> είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί και αν μπορούμε να επιτύχουμε την κατάλληλη πρόοδο. Αλλά υπάρχουν πολλές αναφορές ότι οι μειώσεις εκπομπών που αναφέρονται και πιστοποιούνται δεν αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες χρήσης των οχημάτων αυτών. Πολλές φορές η απόκληση από την πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλη. Και βέβαια οι βιομηχανικοί κύκλοι πολύ λογικά ακολουθούν τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για να γίνει καταμέτρηση των εκπομπών και παίζουν το παιχνίδι αυτό. Όταν το παιχνίδι όμως συνίσταται, όπως μας λένε, συνίσταται σε προσαρμογές στα οχήματα για να μπορέσουν να ε, για να μπορέσει να μειωθεί η αντίσταση στον αέρα του, του αυτοκινήτου, παραγωγός χάρη να ε, γίνονται προσαρμογές στα λάστιχα, να βγαίνουν οι κεραίες, να κλείνουν οι πόρτες ερμητικά, να γίνονται όλα αυτά τα κόλπα για να εξασφαλίζεται ότι θα είναι μεγαλύτερη η ενεργειακή απόδοση του αυτοκινήτου, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται οι υπολογιστέ προς την κατεύθυνση αυτή. Όλα αυτά τα τεχνάσματα χρησιμοποιούνται από τις εταιρείε και αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνουμε την πραγματική ε, τιμή για τις εκπομπές. Κάποιοι μα κοροϊδεύουν με τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι θα χρειαστούν κάποια χρόνια για να έχουμε ένα παγκόσμιο κύκλο δοκιμασιών. Μέχρι τώρα, μέχρι τότε όμως θα πρέπει, όπως ζητήσαμε την Κομισιόν, να υπάρξει μια αναθεώρηση των διαδικασιών δοκιμασίας και θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να καθορίζονται με αυστηρό τρόπο. Αυτό μπορεί να γίνει και μερικές τροπολογίες που έχω καταθέσει, πρέπει όμως να κάνουμε πιο αυστηρό και στεγανό τον τρόπο δοκιμασίας και να εξασφαλίσουμε ότι αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης και έτσι θα έχουμε περιορίσει τα κόλπα και τα τεχνάσματα και θα έχουμε κάνει πιο ρεαλιστική την νομοθεσία μας. Ευχαριστώ κύριε Ντέβις. Είναι παράξενη αυτή η διαδικασία πολλές φορές για τα, τις στα αυτοκίνητα. Κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ πάρα πολύ ενδιαφέρον κύριε Ντέιβις πως ε, Υπενθυμίζετε πως όταν συζητούσαμε την οδηγία πριν από λίγα χρόνια η αυτοκινητοβιομηχανία έφερνε το επιχείρημα πως ε, όλα αυτά τα οποία ζητούσαμε για να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα γεωταχή ή και πιο φιλικά προς το κλίμα ήταν πάρα πολύ ακριβά και δεν ήταν ε, τεχνικώς εφικτά. Χαίρομαι που το διορθώσατε. Ήταν τεχνικώς εφικτά, δεν ήταν πολύ ακριβά και αυτό το μάθημα το ε, παρατηρήσαμε και στις αγορές αυτοκινήτων της Ευρώπης λίγους μήνες μετά. Αναμένω λοιπόν με αγωνία το τι θα γίνει στον επόμενο γύρο ε, συζητήσεων για το εάν δηλαδή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιδείξουμε μεγαλύτερη αντίσταση στα γνωστά επιχειρήματα της βιομηχανίας ή, εάν αυτή τη φορά, θα έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για αυτά τα οποία θέλουμε. Δηλαδή, πρώτον, προστασία των καταναλωτών από μη αποτελεσματικά αυτοκίνητα και πρέπει να προστατευτούν οι καταναλωτές μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγέ πετρελαίου που ήταν πάντα ευρωπαϊκός στόχος και δεν πρέπει να το παραμελούμε. Προστασία του κλίματος. Το φθινόπωρο θα έχουμε τη νέα έκθεση του IPCC και δεν νομίζω πως μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια, ειδικά στον τομέα των μεταφορών, να αμελήσουμε. Επιπλέον, θεωρώ πως στην αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικής βιομηχανίας και καταναλωτών για το ζήτημα της, ε, του μέλλοντος της ευρωπαϊκής αυτοκίνητου βιομηχανίας, το τι δηλαδή θα μπορεί να πουλήσει καλύτερα στο μέλλον η βιομηχανία, νομίζω πως κατά την άποψή μας αυτό είναι πιο αποτελεσματικά και φιλικά προς το κλίμα αυτοκίνητα και όσο πιο καλά τα καταφέρουμε τόσο καλύτερο. Αυτό το οποίο έχουμε τώρα λοιπόν επτάπτωση είναι αντιπαραθέσεις για, τον, για τους στόχους που είναι ήδη στην οδηγία. Δηλαδή μέση όρη διοξείδου του άνθρακα μέχρι το 2020. Αυτά είναι στην παλιά οδηγία. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, κανένας ε, σοβαρός τουλάχιστον δεν τα αμφισβητεί τα 95 γραμμάρια ανά χιλιόμετρα να γίνουν δεσμευτικά. Είναι καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο παρατηρώ μετά την ε, υποβολή της έκθεσης Σούλμα είναι πως δεν αμφισβητείται ο στόχος άμεσα αλλά μέσω των ε, super credits ε, νερώνεται πάρα πολύ. Και αν αυτός είναι ο στόχος του κυρίου Ούλμερ, τότε δεν θεωρώ πως ε, το 95 γραμμάρια κατά μέσο όρο του στόλου της Ευρώπης θα μπορέσουν να επιτευχθούν. Ο κύριος Ούλμερ προτείνει να εγγυηθούμε super credits για μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων, να υπάρξει αυξημένος πολλαπλασιαστής και αυτό το οποίο βρίσκω πιο ξεδιάντροπο προτείνει να υπάρξει και εμπορία αυτών των πιστώσεων. Οπότε ο στόχος που έχουμε για το 2020 θα επιτευχθεί 4-5 χρόνια αργότερα. Και αυτό αντιβαίνει το δεύτερο πράγμα το οποίο λέμε, δηλαδή για το 2025 να έχουμε άλλον δεσμευτικό στόχο. Ο στόχος τον οποίο βρίσκει υπερβολικά φιλόδοξο ο κύριος Ντέιβις, τα 70 γραμμάρια δηλαδή, μπορούν να γίνουν και 60. Ο μακροπρόθεσμος αυτός στόχος είναι σημαντικός γιατί μάθαμε πως τα δεσμευτικά σχέδια των πολιτικών για το πλαίσιο ε, της πολιτικής είναι θετικά. Τώρα, για τον κύκλο δοκιμών. Πέραν της αποτελεσματικότητας των αυτοκινήτων, με την οδηγία αυτή, Εάν έχουμε έναν καλύτερο κύκλο δοκιμών θα προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Οι κύκλοι δοκιμών δεν είναι καλοί, υπάρχουν καλύτερες δυνατότητες και θα έπρεπε να οριστεί το των δυνατών να το συζητήσουμε. Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να βασίζονται στα αποτελέσματα των δοκιμών και αυτό θα γίνει μόνο εάν φροντίσουμε γρήγορα να έχουμε έναν καλύτερο κύκλο δοκιμών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρμς. Μάρτιν Καλάνεν, επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σαν να την έχω ξαναδεί την έκθεση Ντεζαβή για τι εκπομπέ αυτοκινήτων. Πολλές φορές θα συζητήσαμε οι ίδιοι. Καλό που το ξανασυζητάμε. Ευχαριστώ τον Τόμα Σούλμερ. Πολύ καλογραμμένη έκθεση του. Ευπρόσδεκτη απόφασή του να παραμείνει στα πλαίσια τη προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στόχη 130 γραμμάρια από το 2015, 95 γραμμάρια από το 2020 είναι φιλόδοξη, πιστεύω. Στόχοι που η αυτοκινητοβιομηχανία αναγνωρίζει ως επαχθείς, αλλά εφικτούς. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται περί μέσων όρων στόχων για την παραγωγή ε, σε ένα ευρύ φάσμα. Υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος, δύο πλευρές στην εξίσωση. Υποχρεώνουμε τους κατασκευαστές να παράγουν αυτοκίνητα που τηρούν αυτούς τους όρους, απ' την άλλη πλευρά οι καταναλωτές πρέπει να αγοράσουν όμως τα οχήματα που παράγονται σύμφωνα με, αυτά, τα, με αυτές τις τιμές, με αυτά τα όρια. Πολλές από τις αλλαγές που είδαμε πρόσφατα, ε, είδαμε ότι οδήγησε αλλαγές την ζήτηση των αποπλευρά καταναλωτών και η αλλαγή των των καταναλωτών φύγεται στην αύξηση τιμή καυσίμων. Είναι πολύ ανταγωνιστική η κατάσταση που κρατεί. Δεν υπάρχουν πολλοί κατασκευαστέ στην Ευρώπη που κερδίζουν χρήματα. Και δυστυχώ για τον κανονισμό αυτοί που βγάζουν χρήματα είναι αυτοί που βγάζουν τα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, που βγάζουν πολλά καυσάρια. Οι μικροί κατασκευαστέ χάνουν χρήματα και το βλέπουμε γιατί κλείνουν εγκαταστάσει στην Ευρώπη. Πολλά από τα οχήματα ε, εισάγονται από την Κορέα και από αλλού που πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον κανονισμό, αλλά να μην θεωρήσουμε ότι είναι καλό για την ευρωπαϊκή αυτοκίνητη βιομηχανία. Έχουν απώλειες πολλοί κατασκευαστέ. Η αδίποτε ε, μείωση αυτών των ορίων θα είναι μεγάλο σφάλμα, λαμβάνοντα υπόψη και την οικονομική κρίση. Θέλει ο κανονισμό να αναφέρεται στις ε, λεπτομέρειε για την μείωση των στόχων του 2020. Όταν συζητούσαμε αρχικά τον κανονισμό, η ιδέα για να θεσπίσουμε τέτοιου στόχου είναι να δώσουμε μακροχρόνια βεβαιότητα. Το κάναμε αυτό και δεν, έχει, δεν έχουμε λόγο να αλλάξουμε τις κανόνες του παιχνιδιού εν το μέσο της διαδικασίας. Να πω μερικά λόγια για τις λεπτομέρειες τη προτάσεω. Εξαιρέσει κλπ. Καλωσορίζουμε την πρόταση του εισηγητού να διπλασιαστούν οι αρχικέ παρεκκλήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό για τι μικρότερε εταιρείε όπως και οι κατασκευαστές που ε, ε, ε, παράγουν λιγότερα από χίλια αυτοκίνητα επιβατικά το χρόνο. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν κάποιες μικρομεσαίες τέτοιες εταιρείε στην Ευρώπη και δεν επηρεάζουν καθόλου σε σχέση με την παραγωγή. Ελάχιστα οχήματα παράγουν, ελάχιστο ποσοστό και ακόμα μικρότερο ποσοστό οικομπών διοξιδίου του άνθρακος. Άρα πρέπει σύμφωνα με τη γενική τακτική που ακολουθούμε έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να το κάνουμε και εδώ. Το ίδιο ισχύει και την παρέκκληση για διάφορες ε, ειδικέ περιπτώσεις. Παρέκκληση οι κατασκευαστές που παράγουν ειδικά αυτοκίνητα μέχρι το 2020. Θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον χρονισμό υποβολής αιτήσεων για την παρέκκληση κατάλαβε ότι πρέπει να είναι πιο ευέλικτος ο κανονισμός και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις διάφορες ε, ανάγκες των κατασκευαστών και των εμπορευομένων. Τώρα, για τον κύκλο αυτών, τον, τον, κύκλο των δοκιμών, Ανησυχώ λίγο για την πρόταση που αναφέρατε εδώ να εισαχθεί νέα τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών ταχύτερων δυνατών. Οι ισχύοντες στόχοι είναι αυστηροί αλλά εφικτοί και πρέπει να προσέξουμε να μην αλλάξουμε τις κανόνες του παιχνιδιού στο ημίχρονο. Ο κανονισμός ετοιμάστηκε με ένα συγκεκριμένο κύκλο δοκιμών. Αν κινηθούμε προς άλλο κύκλο δοκιμών εντελώς διαφορετικό, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει διαφορετικά αποτελέσματα για διαφορετικού τύπου οχήματα. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε συνετά. Και ίσως το 2020, όταν οι νέοι στόχοι θα καθοριστούν ή λίγο πριν, επανεξετάζουμε το, νέο, το ενδεχόμενο νέο κύκλο δοκιμών, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ αυτό συμβουλεύω. Να μην βιαστούμε να εισάγουμε αμέσω ένα νέο κύκλο. Το ίδιο ισχύει και για την άλλη πρόταση, η καθαριστέρηση τη ρήτη αναθεώρηση για του στόχου μετά το 2020 μέχρι το 2017. Δεν θα πρέπει να δεσμευόμαστε με πιο αυστηρούς στόχου χωρί να έχουμε πλήρη αξιολόγηση συνεπειών. Φαντάζομαι ότι η οικονομική κρίση θα παραμείνει και για τα επόμενα λίγα χρόνια και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στην ευρωπαϊκή παραγωγή και σε σχέση με την παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων θα πρέπει η προσοχή, η σύνεση να είναι βασική, βασικό μας σύνθημα θα πρέπει οι στόχοι να εισάγονται σωστά με σωστή αξιολόγηση συνεπιών, με σωστή μελέτη μακροχρονίων συνεπιών για τη βιομηχανία και να δούμε κατά πόσο εφικτή είναι αυτή η στόχη από πλευρά τεχνολογία. Αυτά και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάλαναν. Ο κύριος Ρώση θα κλείσει τον κατάλογο παρεμβάσεων των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξετίμησα πολύ την παρέμβαση του συναδέλφου Κάλαναν και πλήρως συμμερίζομαι ε, αυτά που είπε. Είπε ο συνάδελφος περίπου κάποια πράγματα σωστά υποστήριξε ότι περνάει η βιομηχανία κρίση και κλείνουν κάποιες μονάδες και μετά υποστηρίζουμε ένα κείμενο που δεν βελτιώνει, δεν βελτιώνει κατά πολύ τις ε, απαγορεύσεις που ζητούνται και του περιορισμού που τίθεται στα Ο καταλαβαίνω ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, διότι δυστυχώ βρίσκεται σε θέση συγκερασμού των διαφορών θέσεων. Κύριε Ρώση, φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα διερμηνία προ τα αγγλικά. Καλώ, μπορείτε να συνεχίσετε. Έλεγα λοιπόν, ο εισηγητή είναι σαφέ ότι έπρεπε να λάβει υπόψη και να συγκεράσει διάφορε τοποθετήσει των ομάδων, όμω έτσι ειλικρινά δεν ελαφρύνει κατά πολύ τι αρνητικέ πιέσει που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστέ αυτοκινήτων. Και από 500 στα 1000 οχήματα να φτάσει το όριο τη εξαιρέσει για τα μικρά αυτοκίνητα, μιλάμε για μια παραγωγή πάρα πολύ μικρή και οι αυτοκινήτων περιορισμένου αριθμού που δίνουν ε, μεγάλα έσοδα, μεγάλη απόδοση στο μικρό κατασκευαστή οικονομική. Και ίσως εκείνα τα οχήματα ε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγάλες επενδύσεις και καινοτομία. Τα μεγάλα εργοστάσια που δίνουν εργασία σε εκατοντάδες χιλιάδες άτομα και που έχουν ε, σαν στυλ παραγωγής το κλασικό αυτοκίνητο, χρήση στο χρηστικό αυτοκίνητο μικρού κόστους που έχει ελάχιστο περιθώριο κέρδους Εκείνε οι μονάδε θα κλείσουν τι εγκαταστάσει, θα παράγουν εκτό Ευρώπη. Και ή κάτι που ήδη συνέβη, Μπορεί να ενδιαφέρονται οι πράσινοι, να, ε, ε, να ενδιαφέρονται εκείνε που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα ποδήλατα. Οι μεγάλες εταιρείε όπω η Fiat, αλλά και άλλε επιχειρήσει. Αναθεώρησαν προς τα κάτω όλες τις συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το τέλος λοιπόν, όχι μόνο αυξήθηκαν οι τιμές των αυτοκινήτων σε σχέση με τα παλιά όρια εκπομπών, αλλά στην πραγματικότητα περιεκόπησαν ε, και οι αμοιβέ και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση την οποία στην Ευρώπη οι εργαζόμενοι αυτού του τομέα για να εργαστούν και για να μην σταλούν στο σπίτι θα πρέπει να πληρώνονται όλο και λιγότερο, αυτή είναι η σωστή ε, προσέγγιση. Πρέπει να τα βάζουμε όλα μαζί. Να λέμε δεν αυξήθηκε, η τιμή, ναι, αλλά μειώθηκαν όμω οι αμοιβέ των εργαζομένων. Αυξάνεται το κόστο τη ζωή και μειώνονται οι αμοιβέ των εργαζομένων στην Ευρώπη. Διότι οι κατασκευαστέ πρέπει να αντιμετωπίσουν παραπάνω δαπάνε όσο εμεί του φορτώνουμε με υποχρεώσει. Συμφωνώ λοιπόν μετά με τον εισηγητή να πρέπει να μεταθέσουμε τη νέα αναθεώρηση μείωση των στόχων. Να ξεκινήσουν συζητήσει. Ε, αργότερα να χρησιμοποιούμε με απλούστερο τρόπο και πιο χρήσιμο τρόπο τις περίφημες πιστώσεις, τα περίφημα credits. Εγώ περίμενα από τον εισηγητή όμως πιο στεναρή προσέγγιση και πιο ευέλικτη, ε, ευέλικτο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των ορίων που είναι πάρα πολύ περιοριστικά. Ελπίζω στο μέλλον εδώ να ξαναμπορέσουμε να συζητήσουμε την όλη κατάσταση, τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη και να μην δυσμονούμε ότι υπάρχει το αυτοκίνητο, αλλά υπάρχει και όλη η αλυσίδα. Ε, Εκείνο που ε, εργάζεται μέσα με την ταπετσαρία, τα χρώματα, βερνίκια, δέρματα, τα ελαστικά κλπ. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο την παραγωγή του αυτοκινήτου αυτού καθεαυτού, αλλά όλη την αγορά και τους εργαζόμενους όλου του τομέα που στρέφεται γύρω από την βιομηχανία. Μιλάμε για μερικά εκατομμύρια εργαζομένους και να μην θεωρήσουμε ότι για να μειώσουμε το κόστος, το τελικό το οχήματος, βλέποντας τις αυξήσεις που επιβάλλουν στην αυτοκινητοβιομηχανία, θα πρέπει να εργάζονται εργαζόμενοι επί όρους σκλαβιάς ή να πληρώνονται πολύ χαμηλά. Να πω και κάτι άλλο ή δυνατόν θα ζητούσα τον εισηγητή τουλάχιστον Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη, αλλά τουλάχιστον απευθύνει έκκληση. Εξή, για χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρικά αυτοκύματα που είναι πολύ καλά για, για τις πόλεις, θα πρέπει τα κράτη-μέλη ε, να ε, ευνοήσουν να δημιουργηθούν διάφορες στήλε φόρτισης των οχημάτων. Διαφορετικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είναι ήδη πιο ακριβά και αν δεν υπάρχει δυνατότητα φόρτωση, οι πολίτε δεν θα αγοράζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν αυτή τη σταθμοί φόρτιση του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρώση. Και τώρα έχω ένα αχανή κατάλογο ομιλητών, 11 ομιλητών που θα λάβουν το λόγο στη συνέχεια και δεν έχουμε αρκετό χρόνο, γι' αυτό προτείνω να έχουμε μοναχά δύο λεπτά ανά ομιλητή. Γκροστέτ, Λάινεν, Λεπάζ, Πανιό, Κράμερ, Λίσε, Βέσλουντ, Σλούτερ, Μαγκάβεν, Φλόρενς και Σέιβερ. Θα ήθελα να κλείσω λοιπόν τον κατάλογο, αν δεν έχετε αντίρρηση, και να δώσω αμέσω το λόγο στην κυρία Γκροστέτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η έκθεση του Τόλμας Ούλμερ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Επικυρώνει τον στόχο των 95 γραμμαρίων μέχρι το 2020 και συμπεριλαμβάνει ρεαλιστικά το θέμα του του κύκλου Υπάρχουν δύο βελτιώσεις που μπορούμε να αναφέρουμε, μία για τα πριμ και δεύτερον για τους κανονισμούς που θα εφαρμοστούν μετά το 2020. Για τα πριμ, η έκθεση Ulmer μας δίνει συγκεκριμένες ε, μορφές κινήτρων στην αυτοκινητοβιομηχανία για να επενδύσουν σε τεχνολογίες που θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Θεωρώ όμως ότι η πρότασή του είναι υπερβολικά πολύπλοκη και δεν είναι ουδέτερη τεχνολογικά, γιατί μονάχα ορισμένε κατηγορίε καινοτόμων αυτοκινήτων θα είναι επιλέξιμε για αυτά τα πρίμα. Εγώ θέλω να καταθέσω μια τροπολογία που να επανεξισορροπήσει αυτή την κατάσταση. Δεύτερον, για την μεταρρύθμιση των κανονισμών μετά το 2020. Θα ήθελα ο κύριο Ούλμερ να μα διευκρινίσει καλύτερα τη θέση του. Λέμε ότι υπάρχει η τροποποίηση αυτή που θα λάβει χώρα μετά το 2020 στην έκθεσή του λέει για τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 το νωρίτερο, το αρχότερο μάλλον, επομένως μπορεί να γίνει πριν από το 2020. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις αυτού του είδους πριν από το 2017. Θα πρέπει να καθορίσουμε καλύτερα τον κύκλο δοκιμασιών πρώτα, να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα, να αξιολογήσουμε τα πρώτα αποτελέσματα και εξάλλου να δούμε και τη διείσδυση στην αγορά των νέων τεχνολογιών, η οποία ακόμα είναι ε, αβέβαια. Γι' αυτό μου φαίνεται ότι είναι πρόωρο να καθορίσουμε πριν από το 2017 τους στόχους μας για επέκεινα του 2020. Αυτά είναι τα δύο σημεία για τα οποία θα καταθέσω τροπολογίες και θα ήθελα να υπάρξουν τροποποίηση στην έκθεση του κ. Ούλμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία ο κύριος ε, ε, Λάινεν, ευχαριστώ. Λέει ο κ. Λάινεν ότι υπάρχει μία παρεξήγηση που πρέπει να ξεπεράσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσει στην αυτοκινητοβιομηχανία ή να την υποχρεώσουμε να αποδεχθεί μειονεκτήματα. Θέλουμε αντίθετα να εξασφαλίσουμε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης θα παίξει ε, κυριαρχικό ρόλο στην ανάπτυξη καινοτομίας και βελτίωσης. Έχουμε ανταγωνιστές από την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και την Κίνα όλο και περισσότερο και βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι είναι παγκόσμιος ο ανταγωνισμός και μόνο τα καλύτερα προϊόντα επιβιώνουν. Η εμπειρία των τελευταίων δέκα ετών κατέδειξε ότι μια φιλόδοξη νομοθεσία μπορεί να βοηθήσει την ευρωπαϊκή αυτοκίνητο βιομηχανία και αντίθετα δεν είναι ένας τρόπος να τις βάζουμε βαρύδια στα πόδια. Πολλοί συνάδελφοι έχουν μιλήσει αν θέλουμε εμεί να δημιουργήσουμε προβλήματα και να επιβάλλουμε κυρώσει στη βιομηχανία. Κάθε άλλο. Όταν το 2008 καθορίστηκαν οι οριακέ τιμέ, υπήρχαν ακριβώ οι ίδιε ανησυχίε και η ίδια αντίσταση που βλέπουμε και σήμερα. Η πραγματικότητα κατέδειξε ότι αυτά βελτίωσαν την απόδοση της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από το αν δεν είχαμε κάνει τέτοιες προδιαγραφές και μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή τεχνολογικών τομών. Όλοι χρησιμοποιούμε αυτοκινήτα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες και κύκλους καύσης που είχαν εφευρεθεί πριν από 100 χρόνια. Έχουν βελτιωθεί εκτοτευσικά, αλλά κατα... καταρχή είναι τεχνολογίες πριν από ένα αιώνα. Και τώρα μιλάμε για τις τεχνολογίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στις επόμενες δεκαετίες και η προσπάθειά μας πρέπει να είναι να έρθουν στην αγορά αυτές οι νέες τεχνολογίες και να βελτιωθεί και η ε, λειτουργία των αυτοκινήτων. Έχουμε την τεχνολογία των κυψελών καύσης, έχουμε τα υβριδικά αυτοκίνητα, την χρήση υδρογόνου ενδεχομένως στο μέλλον και εγώ πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό να θέσουμε φιλόδοξους στόχους, χρειαζόμαστε ε, ένα στόχο και πέρα από το 2020, το ξέρουν οι βιομηχανικοί κύκλοι και εν μέρει αναμένουν να θέσουμε εμείς κάποιους τέτοιους στόχους. Για τα super credits και τα συστήματα κινήτρων, ναι, αλλά όχι για να αποδυναμώσουμε τους στόχους. Δεν πρέπει να έχουμε ένα παράγοντα τρία, γιατί αυτό ουσιαστικά ε, αποδυναμώνει και αλλοιώνει το στόχο του 95 γραμμαρίων. Λεπάζου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ακολουθώ αυτά που είπε ο Γιολάινεν προηγουμένω. Το ουσιαστικό εδώ είναι να εξασφαλίσουμε και μια βιώσιμη μορφή οικονομικής ανάπτυξης για, τον στόχο, για την αυτοκινητοβιομηχανία και να επιτύχουμε συγχρόνως και τους στόχους μείωσης των εκπομπών. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να θεσπίσουμε στόχους οι οποίοι θα είναι φιλόσοφοι, φιλόδοξοι συγγνώμη, και οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις μας. Δηλαδή να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο, ο συν, συντελεστής κατανομής των προσπαθειών να ανταποκρίνεται στους κανόνες ανταγωνισμών μεταξύ των επιχειρήσεων. Γι' αυτό εγώ υποστήριζω περισσότερο να χρησιμοποιούμε άλλους ε, άλλα κριτήρια και όχι τα κριτήρια της μάζας που έχει η Κομισιόν. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο καθορίσουμε από τώρα στόχους για το επέκεινα του 2020, όπως λέγαμε και χθε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει η βιομηχανία τι επίκειται, ποια θα είναι η πορεία του μέλλοντος. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε την ρήτρα επανεξέτασης για το 2017. Για τους μηχανισμούς τώρα της καινοτομίας, δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε στευλός και να καταλήξουμε σε αποτελέσματα αντίμαχα αυτών που θέλουμε να έχουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια και τον πραγματικό χαρακτήρα. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε τα πιο ε, πρόσφατα στοιχεία του 2009 και του 2006 και να εξασφαλίσουμε ότι οι δοκιμασίες θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην πραγματική χρήση, όχι μόνο για να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών, αλλά για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το βασικό μας στόχο που είναι η μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεπάς. Ο κύριος Πανιού έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι σημαντικό στα πλαίσια αυτής της προτάσεως κανονισμού να, που, να έχουμε υπόψη ότι αυτό που συζητούμε και αυτό που θα προτείνουμε δεν αποτελεί κύρωση για την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά ένα όφελος πλεονέκτημα που θα επιτρέψει στην αυτοκινητοβιομηχανία όχι μόνο να προστατεύσει και να όλους τους καταναλωτές και να καταπολεμήσει καλύτερα τη θέρμανση λόγω της αλλαγής του κλίματος, αλλά θα επιτραπεί επίσης στον τομέα να βρει λύσεις και έτσι θα μπορούν αύριο να κατασκευάζουν καθαρά αυτοκίνητα. Είναι σημαντικότατο Επίσης αυτή η πρόταση κανονισμού να επιτρέπει ισότιμη αντιμετώπιση, ισότητα για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και κυρίως μετά το 2020 κάποιες παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση θέλουμε για το 2020 η κατανομή της προσπάθειας μεταξύ κατασκευαστών να στηρίζεται αυτό που είπε η κυρία Λεπάζ σε αρχή χρησιμότητας και ίχνους στο έδαφος και ο συντελεστής ε, κατανομής της προσπάθειας να υπολογίζεται βάση διαθεσίμων στοιχείων ε, από πλευράς βιομηχανίας τα πιο πρόσφατα στοιχεία ε, εκείνα του 2009 και του 2006. Μετά το 2020 θέλουμε ταυτόσιμος στόχος για το διοξείδιο του άνθρακος να ισχύει για όλους τους κατασκευαστές και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει ρήτρα αναθεώρησης το 2014 και όχι το 2017. Και κλείνοντας, δεν είμαι υπέρ της παράτασης των αυτών των, ε, των ε, αυτών των κινήτρων διότι κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε το μηχανισμό μας ε, και μάλιστα στη συνάρτηση με τους στόχους που έχουμε καθορίσει για το 2020. Ευχαριστώ πολύ. Κράμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που έχει υποβάλει μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Θα αναφερθώ σε όλα τα επιχειρήματα που είπε ο ίδιο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Θα πω κάτι το οποίο ισχύει για τα ελαφρά φορτηγά, τα οποία παρακολουθώ εγώ. Δεν υπάρχει αυτόματη σχέση μεταξύ χαμηλών εκπομπών και εμπορικής επιτυχίας. Γιατί όσοι θεωρούν πως βοηθάνε την βιομηχανία έτσι πρέπει να το ξέρουν. Το αντίθετο συμβαίνει μάλιστα άμα δείτε. Όσοι εκπέμπουν περισσότερα ε, πουλάνε και, και περισσότερα αυτοκίνητα. Άρα η επιτυχία δεν προέρχεται από τα μικρά αυτοκίνητα αλλά από τον τομέα των πολυτελών αυτοκινήτων. Και βεβαίως έχουμε ήδη φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων της φυσικής τουλάχιστον να μιλάμε για κινητήρες εσωτερικής καύσης και πράγματι εφευρέθηκε πριν από 100 χρόνια ο κινητήρας εσωτερικής καύσης μα και ο κινητήρας ε, ο ηλεκτρικός εφευρέθηκε πριν από έναν αιώνα και όλα τα πειράματα είχαν αποτύχει για λόγους ε, τεχνολογικούς, ε, οικονομικούς και δεν βλέπω μεγάλα επιχειρήματα για αυτό το οποίο λέτε ότι είμαστε ενώπιον μια μεγάλη τεχνολογική αλλαγή. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Μπορεί να είναι το φυσικό αέριο, μπορεί να είναι μια άλλη ε, τεχνολογία, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτά τα οποία ε, φανταζόμαστε για μετά το 2020. Ό,τι γράψουμε εμείς σήμερα είναι πολιτικά νούμερα, έτσι, είναι εκτιμήσεις. Μπορούμε να γράψουμε 60-70 ό,τι θέλουμε, ένα νούμερο όσο πιο φιλόδοξο τόσο πιο καλύτερο. Αλλά δεν είναι σαφές το τι θα γίνει, ε, το πώς θα επιτευχθούν επίσης αυτά με τη σημερινή τεχνολογία. Με όλα όσα συζητάμε επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε πως από όλε τι νομοθεσίες που υπάρχουν παγκοσμίω, όλα αυτά ρυθμίζονται βεβαίως, ε, έχουμε εμεί την πιο φιλόδοξη. Την πιο φιλόδοξη παγκοσμίω από ΙΠΑ, Καλιφόρνια, Κορέα. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Και υπάρχει ένα όλο ε, και μικρότερο όριο, μια λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ κινήτρου και τιμωρίας πλέον. Και άρα ε, αυτά τα οποία προτείνει ο κύριος ε, Ούλμερ νομίζω είναι σωστά. Κατά την Ευχαριστώ. Πέτερ Λίζε. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Τόμας Ούλμερ για το σχέδιο έκθεσης. Είναι μια πραγματικά καλή βάση και πολλά πράγματα μπορούμε να τα στηρίξουμε. Εγώ είμαι υπέρ του να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τα super credits για να προωθήσουμε την καινοτομία. Βεβαίως δεν ξέρω το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος εάν ορίσουμε κάποιο όριο ή κάτι άλλο. Δύο σημεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πρώτον, ο κύκλος δοκιμών. Χθες μιλήσαμε πάρα πολύ για το ε, κρέας των αλόγων. Για να κάνω μια παρομοίωση. Ε, είναι όχι μόνο σαν να βάζαμε στα λαζάνια κρέας αλόγου, αλλά να το εγκρίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύκλο δοκιμών δεν περιγράφει σωστά την κατάσταση. Όποιος έχει οδηγήσει αυτοκίνητο το ξέρει. Ξέρει πω δεν πετυχαίνει ποτέ. Αυτού του στόχου μπορεί να οδηγάει όσο προσεκτικά θέλει, αλλά δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Και απογοητεύονται και εξαπατώνται οι καταναλωτέ. Και όπω είπα είναι μία μικρή ε, απάτη ε, είναι κάτι το ε, εκνευριστικό γιατί το συζητάμε χρόνια και δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, γιατί μετά από 15 χρόνια σε διεθνέ επίπεδο δεν γίνεται τίποτα. Και όπως είπα είναι παραπλάνηση των καταναλωτών. Τελευταίο, ε, επόμενο σημείο, μακροπρόθεσμο στόχος. Εγώ είμαι υπέρ του να γράψουμε κάτι. Όχι πολύ φιλόδοξο. Αλλά δεν θέλω να ζήσω αυτό το οποίο έχουμε ζήσει πολλές φορές. Δηλαδή υπήρξε πριν από πολλά χρόνια η εθελοντική συμφωνία, δεν τηρήθηκε και λέμε θέμε μόνο να τηρηθεί η εθελοντική συμφωνία σε ένα νόμο, άμα τώρα είναι αργά. Και θα επαναληφθεί αυτή η υπόθεση αν δεν κάνουμε κάτι τώρα. Γιατί ε, αν πούμε τώρα πως ναι είναι πολύ αργά, σε πέντε χρόνια πάλι πολύ αργά θα είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να θέσουμε ένα στόχο ρεαλιστικό, αλλά όπως είπα ε, κάτι που κάποτε πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ Βέστλοντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι εύκολο να περάσουμε σε τεχνική συζήτηση όταν μιλάμε για αυτή την τεχνολογία, αλλά νομίζω πως πρέπει να θυμόμαστε το τι κάνουμε εδώ πέρα. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνο για ένα μεγάλο ποσοστό, οπότε αυτός ο τομέας πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να οδηγάμε αυτοκίνητα, πρέπει κάθε αυτοκίνητο να εκπέμπει λιγότερο, αλλιώς δεν θα γίνεται. Νομίζω λοιπόν πως τα 95 γραμμάρια ήταν μια από τις πιο συναρπαστικές αποφάσεις ε, που είχαν ληφθεί ποτέ. Και η αυτοκινητομηχανία μας είπε πως δεν θα γίνει ποτέ, μια χαρά έγινε και είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θεωρώ πως πρέπει να θέσουμε μακροπρόθεσμους στόχους. Αντιλαμβάνομαι τα επιχειρηματά που ακούμε, πως ο κύκλος δοκιμών πρέπει να αναθεωρηθεί, αλλά νομίζω πως πρέπει να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο ενδεικτικό στόχο που μπορεί μετά να αναθεωρηθεί με βάση τον νέο κύκλο δοκιμών. Δεν έχει νόημα να μην θέσουμε ε, μακροπρόθεσμο στόχο και να το κάνουμε όταν θα έχουμε νέο κύκλο δοκιμών, θα μας πει η αυτοκινητομηχανία τότε μα δεν υπάρχει χρόνος. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι σημαντικός για τους κατασκευαστές και για εμάς που πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να προστατεύσουμε την εξαίρεση ε, για τους μικρούς, ε, να διατηρήσουμε εξαίρεση για τους μικρούς κατασκευαστέ. Υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι για να πει κανείς πως ε, ένα μεγάλο αυτοκίνητο ε, εκπέμπει περισσότερο από ένα μικρό. Αλλά αν θέλει κανείς να αγοράσει ένα φοβερό σπόρο αυτοκίνητο πρέπει να πληρώνει για τις εκπομπές. Γιατί να εξαιρεθεί. Yeah. I say the same thing here. Και εγώ τα λέω τα ίδια πράγματα. Αυτοί που θέλουν να πουλήσουν αυτοκίνητα στο μέλλον θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με την ε, χρήση ενέργειας. Στον τρίτο κόσμο, στην Ινδία, στην Αφρική δεν μπορεί κανείς να αγοράσει αυτοκίνητα που εκπέμπουν τόσο πολλούς ρήπους και καταλαλώνουν τόσο πολύ ε, πολλά καύσιμα. Ο στόχος του 2015 έχει επιτευχθεί ήδη το 2011. Είμαστε μονάχα λίγα γραμμάρια μακριά γι' αυτό. Επομένως νομίζω ο μόνος λογικός δρόμος είναι να προχωρήσουμε προς πιο ε, αυστηρά πρότυπα. Γιατί Εάν δεν το κάνουμε εδώ, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό για την αυτοκινητοβιομηχανία μας. Όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη είναι έτοιμες να φτάσουν τους στόχους αυτούς. Στην Ιταλία έχουν κατέβει ήδη κάτω από το 130 γραμμάρια. Και τα 95 είναι πολλά. Χρειαζόμαστε ένα πιο στεναρό στόχο για το 2025. 60 γραμμάρια <clears throat> είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό και για τους περισσότερους κατασκευαστές, ακόμα και χωρίς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και γιατί να έχουμε super credits για χαλαρά πρότυπα. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Δεν πρόκειται να βελτιώσει την τεχνολογία. Αυτό το οποίο οδηγεί τις τεχνολογίες είναι τα αυστηρά πρότυπα. Να έχουμε υπερπιστώσεις super credits για να διατηρήσουμε χαλαρά standards, αυτό δεν έχει νόημα. Αν θέλετε ένα σύστημα καινοτομία στην Ευρώπη θα πρέπει να ακολουθήσετε πιο αυστηρές απαιτήσει και αν θυμηθούμε το σκάνδαλο του αλογίσιου κρέας, κρέατος. Γιατί να επιτρέψουμε ένα κύκλο δοκιμασιών όπου είναι μία απάτη. Κα... Κοροϊδεύουμε όλους αυτούς που αγοράζουν αυτοκίνητα στην Ευρώπη. 20-30 περισσότερο εκπομπές είναι στην πραγματικότητα αυτές που έχει να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής εναντί των κύκλων δοκιμών. Και τώρα λέμε να καθυστερήσουμε την εφαρμογή ενό νέου κύκλου δοκιμών μέχρι το 2020. Γιατί, 21, γιατί να το καθυστερήσουμε. Θα πρέπει από τώρα να έχουμε ένα νέο κύκλο και να προσαρμόσουμε τα πρότυπα σε αυτό τον κύκλο. Αυτό είναι η μόνη λογική προσέγγιση. Ευχαριστώ, Πάουλ. Η Λίντα Μαγκέβεν Και εγώ θα μιλήσω. Υποστηρίζω όλους όσους είπαν ότι θέλουμε κάποιο στόχο μετά το 2020. Η βιομηχανία πάντα παραπονιούται και λέει ότι δεν έχει χρόνο για στόχους, ας μην καθυστερούμε τον καθορισμό στόχων, ώστε να μην μας λένε μετά σε τέσσερα χρόνια να αργά να καθορίσουμε άλλους στόχους. Ξέρουν την τεχνολογία οι εταιρείε, ξέρουν τι είναι εφικτό, το είπε και ο Τζον Λάινον. Μπορούμε να θέσουμε νέους στόχους. Δεύτερον, συμφωνώ με όλους με αυτά που είπε ο Πίτερ Λίζε και ο συνάδελφος Μάριο Περίλιο και άλλοι για τον κύκλο των δοκιμών. Α σκεφτούμε τι κάνει ο καταναλωτή. Εγώ ήθελα να αγοράσω ένα καινούριο αυτοκίνητο το ψαχνά, προσπαθούσα να συγκρίνω εκπομπέ άνθρακο των διαφόρων χημάτων. Είναι η αιωνία δύνατο να καταλάβει ο καταναλωτή, διότι βλέπει κανεί τα στοιχεία που δίνει από του πολιτέ. Συγκρίνει τα στοιχεία με του εμπειρογνώμονε και άλλου που λένε όχι στον πραγματικό κόσμο. Σου λένε αυτό το όχημα βγάζει τρία γραμμάρια, τέσσερα γραμμάρια παραπάνω. Ο κόσμο πώ να έχει εμπιστοσύνη στο σύστημα και αν δεν έχει εμπιστοσύνη, γιατί να πληρώσει και κάτι παραπάνω για να αγοράσει αυτά τα αυτοκίνητα και τώρα πληρώνουν πολλά περισσότερα. Κοίταξα τις τιμές. Τις συνέκρινα με τιμές ηλεκτρικών και υβριδικών στη ΣΥΠΑ. Πληρώνουμε πολύ περισσότερα στην Ευρώπη για αυτού του είδους τα οχήματα. Αν θέλουμε ο κόσμος να τα αγοράζει θα πρέπει να ξέρουν και την αλήθεια. Είναι κατεπήγον ζήτημα και δεν μπορεί να καθυστερήσει και να το αφήσουμε και να το κρύψουμε και να το θάψουμε. Ευχαριστώ κυρία Μαγκόβαν. Ο Καλ Χάιντς Φλόρεντς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Τόμας Ούλμερ ειδικά για το ότι ε, μας ανέφεραν ο κύριος Κάλλαν και ο κύριος Ρώση διάφορες ιστορίες. Ναι, εγώ θεωρώ πως είναι καλή εκτίση πηγαίνει ε, σωστή κατεύθυνση. Θέλω να εξηγήσω τώρα ξανά το όνειρο των 95 ε, γραμμαρίων. Ο κύριος Κάλλαν βεβαίως λυπάται γιατί εμείς θέλαμε κάτι πολύ αυστηρότερο, αλλά τελικά προέκυψαν τα 95 γραμμάρια από τη διαδικασία της συνδιαλλαγής, γιατί κάποιες χώρες ε, ήθελαν να στηρίξουν ε, τον ε, κλάδο. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ θεωρώ πως θα έχουμε ένα παγκόσμιο ανταγωνισμό και θα κινδυνεύσει η αυτοκινητομηχανία στην Ευρώπη. Δηλαδή οι χώρες οι οποίες είναι αποτελεσματικές θα κερδίσουν εκεί πέρα. Κοιτάξτε λοιπόν, λόγω του χρόνου σύντομα. Εγώ ήμουν υπέρ των ε, super ε, credits Γι' αυτό ε, προτείνω γύρω από τα super credits να θέσουμε έναν στόχο διαφορετικό. Δεν είναι δυνατόν να σημαίνει πως ε, έχει κανείς δύο γραμμάρια παραπάνω. Για, έτσι για να έχει κάποιο δώρο. Μάλιστα και η Ένωση των Αυτοκινητομηχανίων δεν είναι τόσο πολύ κατά. Μακροπρόθεσμα συμφωνώ για να έχουμε στόχο, αλλά όχι ε, αυτό το παγιωμένο, τυχαίο ε, τα 95 γραμμάρια. Να κάνουμε ένα γραμμά, ένα διάδρομο, εάν θέλετε μεταξύ δύο αριθμών. Και σα εγγυώμαι πω περισσότερε εταιρείε θα είναι στο αυστηρότερο άκρο. Η Fiat ήδη τα κάνει σήμερα. Μπορεί να επιτύχει αυτό τον στόχο. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο για τον ε, κύκλο δοκιμών. Αν ε, εσεί όλοι που υπερασπίζετε τον κύκλο δοκιμών θέλετε να εξηγήσετε στα παιδιά σα αυτό το πράγμα, αν το λέγατε στα παιδιά σα, «Μάρε μπαμπά, πού δουλεύει, τι μπούρδε είναι αυτέ. Thank Ευχαριστώ κύριε Φλόρενς, σας έδωσα και άλλο χρόνο για να πέσετε τις τελευταίες δύο φράσεις σας. Ο κύριος Σέιμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προστασία του κλίματος πρέπει να γίνεται όσο δυνατόν πιο οικονομικά και δεύτερον θεωρώ πως η αυτοκινητομηχανία μας βρίσκεται και σε έναν διεθνή ανταγωνισμό. Σημαντικό είναι λοιπόν να έχουμε κατά νου πως τεχνολογικά σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερες οι δυνατότητες. Δεν το συζητάμε αυτό. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ε, είναι πάνω από 100 ετών. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε την πραγματικότητα. Δεν έχει νόημα τώρα να θεωρούμε πως με κάποιες διατάξεις εμείς ε, θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε την ε, τεχνολογία και το που θα κινηθεί. Θέλουμε λοιπόν αποτελεσματικότητα, στα καύσιμα, θέλουμε ε, λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα ή θέλουμε πιο αθόρυβα αυτοκίνητα. Όλα αυτά μαζί δεν πάνε γιατί καμιά φορά το ένα πάει αντίθετα από το άλλο. Πρέπει λοιπόν να ξεχαρίσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμα. Και το βασικό είναι πως ε, οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι για να πούν οι εταιρείε εμένα με ενδιαφέρει αυτή η τεχνολογική λύση και η ιδέα των super credits ε, έχει κάποιο νόημα. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε οπωσδήποτε τον ε, κύκλο δοκιμών και τις τιμές. Μα, αν αλλάξουμε τον κύκλο δοκιμών πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τις τιμές που ορίζουμε. Και σας παρακαλώ μην ξεχνάμε το εξής. Δεν ισχύει το ότι όλα αυτά δεν έχουν κόστος. Είναι απλά λάθος. Τα πληρώνει ο καταναλωτής πρέπει να το σκεφτούμε αυτό όταν τα κάνουμε πιο αυστηρά. Θα, ε, πρέπει να το σκεφτούμε ότι γίνεται ακριβότερα τα αυτοκίνητα τα ευρωπαϊκά και για τους Ευρωπαίους. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μία μέση οδό, ναι, προστασία του κλίματος, ναι, καινοτομία, αλλά και την πλευρά του κόστους. Δεν μπορεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής να πληρώνει πολύ περισσότερο για το αυτοκίνητό του από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σέμπερ. Τελευταίος που θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά είναι η κυρία Ακόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι τελευταία. Πολλά ήδη υπόθηκαν. Δεν θα τα επαναλάβω όλα. Μακροπρόθεσμη μακροπρόθεσμοι στόχοι και το σύστημα των δοκιμών λοιπά, Όλα αυτά έχουν υποθεί. Νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Έλμερ είναι μια έκθεση που επιτρέπει σωστή ισορροπία, καλή ισορροπία μεταξύ προστασία του περιβάλλοντο από τη μια με την προστασία τη βιομηχανίας από την άλλη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η βιομηχανία μα, η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει μεγάλες συνέπειες ε, για μερικέ από αυτέ τι αυτοκινητοβιομηχανίε και θα πρέπει να έχουμε υπεύθυνη νομοθεσία. Όπω είπε ο Ρίτσαρ Σέμπερ, κάποιες προδιαγραφές αλλεπάλληλες επιβαρύνουν και δυσκολεύουν την βιομηχανία, την εμποδίζουν να μπει στην καινοτομία, διότι δημιουργούμε μία αστάθεια νομική και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν βελτιώσεις που μπορούν ε, να επιτευθούν και συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του κυρίου εισηγητού. Θέλουμε να μειώσουμε τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου και η προστασία των αποστατεύσεων των περιβάλλων, περιβάλλον, από τη μια και από την άλλη προστατεύσουμε και την αυτοκινητοβιομηχανία μα και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε ποτέ. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κόνη, ήξερα ότι στην αυτοκινητοβιομηχανία μιλάτε για υποδύναμη, αλλά βρήκαμε τώρα και ε, συσχετισμό μεταξύ αυτοκινήτων και κρέατο ε, ύπου. Θα ήθελα να ξέρω τι έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτό. Κύριε Όουεν, να σα δώσω το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε αυτό που ήθελα. Μιλούσαμε για υποδύναμη ε, και μιλούσαμε και για αλογίσιο κρέας κλπ. Ε, χαίρομαι που ε, το θέσατε έτσι το ζήτημα. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Ούλμερ για την πλήρη έκθεσή του και θα ήθελα όπως και ο κύριος Ντέιβεν συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία. Θα θυμόσαστε τις εθελοντικές συμφωνίες που εφαρμόστηκαν πριν μερικά χρόνια και δεν έδωσαν αποτελέσματα αλλά και με τη δεσμευτική νομοθεσία μείωσε με επιτυχία τις εκπομπές από 160 σε 135 γραμμάρια το 2011 η αυτοκινητοβιομηχανία και είναι καθοδόν προς επίτευξη στόχο στόχου 130 γραμμαρίων πριν το 2015. Ε, και γι' αυτό εμείς έχουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά κάποιες από τις προτάσεις του κυρίου Ούλμερ. Βασικά όσον αφορά τα super credits, Άκουσα πολύ κόσμο να λέει ότι πρέπει να διατηρήσουμε το στόχο των 130 γραμμαρίων και τα 95 γραμμάρια να τα κρατήσουμε και να τα μειώσουμε αυτά τα όρια. Να τα αποδυναμώσουμε, αποδυναμώσουμε του περιορισμού. Αλλά δεν, χρει... δεν νομίζω ότι τα super credits οδηγούν σε μείωση αυτών των στόχων. Τα 130 γραμμάρια για το 2015 ε, θα πληγεί διότι θα γίνει εμπόριο μεταξύ 2015-2016, ε, θεσπίζονται και νέα κριτήρια για τον υπολογισμό των super credit για αυτή την περίοδο, 40 χιλιόμετρα ε, με ηλεκτροκίνηση. Αλλάζει λοιπόν, ε, αλλάζουν οι όροι για την αυτοκινητομηχανία και μειώνεται η βεβαιότητα. Τα 95 γραμμάρια, ο στόχος και αυτός επηρεάζεται κατά 15% μέχρι 109 γραμμάρια επιτρέποντας αυτή την προβλεπόμενη συναλλαγή. Και δεν είναι καλή λύση. Ε, το αποθεματικό. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι κατά την περίοδο μεταξύ 2020 και 2030 αν τα κράτη-μέλη 50% ο στόχος του 50% επιτευθεί θα έχουμε άλλα, άλλα 120 εκατομμύρια τόνου διοξιδίου του άνθρακου που θα ελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα αυτή την περίοδο. Πολλοί μίλησαν για τον κύκλο των δοκιμών και θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι εδώ. Τι προτείναμε. Αν εισαχθεί νέο κύκλο, θα προσαρμόζαμε τα στοιχεία δεόντω. Θα βρίσκαμε κάποιου σχετισμούς. Και έτσι ο στόχο των 95 ε, γραμμαρίου να μην γίνει αυστηρότερος. Ήμασταν πολύ ανοιχτοί και διαφανεί στην πρότασή μα η θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 ε, να δώσει το WLBT και θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε πολύ Λοιπόν, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το σύστημα διότι είναι παλιό το άλλο και επικαιροποίηση αυτού θα μπορούσε να οδηγήσει στην αλλαγή το νέο ευρωπαϊκό, το κύκλο οδήγηση και λοιπά να την υπόψη ε, και δεν θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση οτιδήποτε κατασκευαστή. Λοιπόν, οι παρεκκλήσει για το μικρό όγκο που ανέφεραν διάφοροι ε, και η έκθεση προτείνει μία αύξηση των δοκιμών από 500 σε 1000 οχήματα ε, εγώ κατανοώ, θέλω να μειώσουμε το βάρος που στο οποίο υπόκεινται μικρές εταιρείε, αλλά δεν είναι τόσο μικρές αυτές οι εταιρείε και αυξάνοντας σε χίλια αυτοκίνητα βγάλουμε ε, την Αλπίνα εκτός μάχης στην ε, Γερμανία ή την Λότους στο Ηνωμένο Βασίλειο από το πεδίο εφαρμογή και πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς τι κάνουμε. Λοιπόν, όσον αφορά την αναθεώρηση ε, ακούσαμε όλοι ότι χρειάζεται να υπάρχει ε, σχεδιασμός, ε, να υπάρχει βεβαιότητα στον σχεδιασμό και θέλουμε να δώσουμε αυτή την να δώσουμε και χρόνο στους, στις εταιρείε να προσαρμόσουν τους τόλους. Χρειάζεται 5-6 χρόνια να αλλάξει ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου, 10 χρόνια για να αλλάξει ο σχεδιασμός κινητήρων. Θα πρέπει λοιπόν τώρα το ταχύτερο δυνατόν μετά την εξολόγηση αντικτύπων να καθορίσουμε κάποιους στόχους για το περίοδο μετά το 2020. Και πρόθεσή μας είναι ταχύτερο δυνατόν να δώσουμε ανακοίνωση ούτως ώστε να μπορούμε να συγκεράσουμε τις ιδέες και να ξεκινήσουμε τις προσπάθειες για την αναθεώρηση του 2014 και δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε όσον αφορά το θέμα, αν είναι αυτό δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Owen. Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω τον εισηγητή κύριε Ölmer για να κλείσει την συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να κάνω μια σύντομη σύνοψη. Εγώ δεν θεωρώ ότι η πρότασή μου αποτελεί κυρώσεις εναντίον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αντίθετα είναι ένα σύστημα κινήτρων το οποίο μπορεί να τις βοηθήσει να αναβαθμίσουν την τεχνολογία που χρησιμοποιούν για τα αυτοκίνητά τους. Όταν μιλάμε για τα super credits, εγώ νομίζω ότι είναι σαφής η λογική που ακολουθούμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή 85 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ευρώπη και έχουμε μονάχα 12 περίπου εκατομμύρια τα οποία τίθενται στην κυκλοφορία κάθε χρόνο. Τα super credits ουσιαστικά θα αφορούν μονάχα το ένα χιλιοστό αυτών των αυτοκινήτων. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να έχουμε ένα σύστημα, ένα μικρό σύστημα κινήτρων προς την κατεύθυνση της βιομηχανίας ώστε να υπάρξει μια ταχύτερη και πιο εντατική και πιο φιλόδοξη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που θα μειώσουν αν θέλουμε να έχουμε μια πιο μεγάλη πώληση κατά 10% παγκόσμιο χάρη στην ε, πώληση αυτοκινήτων, νέων αυτοκινήτων, είναι χρήσιμα αυτά τα κριτήρια για να μπορέσουν να προωθήσουν τη χρήση αυτοκινήτων που έχουν καλύτερες και όχι χειρότερες τιμές εκπομπών. Ήδη έχουμε πάρει μια απόφαση για το ETS. που ουσιαστικά σημαίνει μια μείωση των τιμών των ε, πιστοποιητικών για τις εταιρείες. Τώρα μιλήσαμε για τον κύκλο δοκιμών, αυτό βέβαια δεν είναι ένα πρόβλημα. Η Κομισιό μας έχει διαβεβαιώσει ότι μπορεί να λάβει υπόψη ένα παράγοντα προσαρμογής ώστε να παραμείνουν μέσα στα πλαίσια της ε, πραγματικότητος οι δοκιμές αυτές. και να μπορεί να εξηγήσει τον καταναλωτή αν θεωρεί ότι καταναλώνει πάρα πολύ το όχημα το οποίο έχει αγοράσει. Πιστεύουμε ότι πολλά από αυτά μπορούν να εφαρμοστούν, όχι όμως πλήρως. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα κοινό στόχο μετά από το 2020, και εγώ πιστεύω ότι αυτός θα πρέπει να είναι ένας φιλόδοξος στόχος για όλους και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια οριακή τιμή για το διοξείδιο του άνθρακος που επέμπεται ή το αντίστοιχό του Εάν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ισοδύναμο διοξιδίου του άνθρακος το οποίο εκλείεται από τη διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής για τα ηλεκτρικά αυτά αυτοκίνητα. Για αυτά, αυτά λοιπόν θα ήθελα να πω και σας ευχαριστώ για όλες τις συνεισφορές και προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της συζήτησης. πολύ κύριε Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τα νέα επιβατικά οχήματα. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι την επόμενη Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου. Θα εξεταστούν οι τροπολογίες συνεδρία τη Επιτροπής τη 20-21 Μαρτίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 24-25 Απριλίου και ε, δεικτικό σχεδιασμό στην Ολομέλεια είναι Ιούνιο φέτο. Προχωρούμε τώρα στο σημείο 10. Αφορά κλινικές δοκιμές. Όποιος θέλει να αποχωρήσει από την αίθουσα, παρακαλώ ας αποχωρήσει γρήγορα και ήσυχα. Δίνω στην εισηγήτρια την κυρία Βίλμοντ το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Προεδρία του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους σκιώδεις συζητητές. Ήταν έξοχη η συνεργασία μας μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αληθεύει το ότι ήθελαν όλοι να πετύχουμε το ταχύτερο δυνατόν καλή συμφωνία πάνω σε ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν ότι η παρούσα νομοθεσία όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές χρήζει επιγόντως αναθεωρήσεως. Είδαμε μεγάλη μείωση των κλινικών δοκιμών που, που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, που διενεργούνται στην Ευρώπη. Σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, μπορείτε να αποχωρήσετε ήσυχα από την αίθουσα, διότι συνεχίζεται η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το 2007 μέχρι το 2011 ο αριθμός των δοκιμών που διενεργήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 25% περίπου, κατά τον τέταρτο, και αυτό έχει σοβαρότερες οικονομικές συνέπειες, αλλά παρεμποδίζει και την πρόοδο της ιατρικής εις των ασθενών. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι η Ευρώπη ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο στην έρευνα. Επίση όμω θα πρέπει να εξασφαλίζουμε το ότι προωθούμε και την ακαδημαϊκή έρευνα και ενθαρρύνουμε και την ανάπτυξη φαρμάκων για σπάνιε ασθένειε. Ταυτόχρονα πρέπει να ηγείται η Ευρώπη και στην ασφάλεια των ασθενών και στη διαφάνεια προ όφελο τη εμπιστοσύνη του κοινού ε, και της ε, σωστής ανάπτυξης της επιστήμης. Καλωσορίζω πολλά από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρώτα απ' όλα θα ασχοληθώ με αυτά τα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό και όχι η οδηγία. Νομίζω ότι το αμάγαλμα των διαφόρων νομοθεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε σε δύσκολε ε, δυσνορικές δοκιμέ και δαπανηρέ. και είναι πάρα πολύ δύσκολο για εκείνου που ασχολούνται με σπάνιε ασθένειε, όπου υπάρχει μικρό πληθυσμό των ασθενών άρα θα πρέπει να γίνεται επεξεργασία διασυνοριακά. Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα για την έγκριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πάρα πολλά από τι ρυθμιστικέ αρχέ, τις διοντολογικές αρχές ε, διοντολογικές και τους χορηγούς ε, και γίνονται πιο δαπανηρές οι δοκιμές όσο χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Τα χρονοδιαγράμματα είναι άκρο φιλόδοξα, αλλά είναι εφικτά και βασίζονται στι βέλτιστε πρακτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιε ανησυχίε όσον αφορά τι προθεσμίε που θεωρούνται πάρα σύντομε σύντομες, αλλά πολλά κράτη-μέλη που θέλουν να παρατείνουν αυτά τα χρονοδιάγραμματα Θέλω τελικά όμως να καταλήξουμε σε καλή συμβαστική λύση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε ισχυρή διαπραγματευτική θέση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ε, ένα, μια από ιδέες είναι της ε, πύλης στο, στο, στο διαδίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε θα μπορεί να είναι πιο εύκολη η αδειοδότηση και η έγκριση και θα είναι κάτι επωφελές για αυτούς που ασχολούνται με σπάνιες ασθένειες. Και η έννοια της μικρής, ε, των, παρε, των δοκιμών χαμηλής παρέμβασης ε, που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία γιατί θα είναι μικρότερος ο κίνδυνος σοφά τις δοκιμές. Μειώνεται η γραφειοκρατία μένα από τη μία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη ε, την ασφάλεια των ασθενών και είναι μέγιστη προτεραιότητα. Πρότεινε τη συμμετοχή των ασθενών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση των κλινικών δοκιμών, το υποστηρίζω αυτό. Ε, Όμω θέλω αυτοί οι ασθενεί ε, να είναι έμπειροι και να γνωρίζουν και η συμμετοχή του να μην ειδωθεί σαν κάτι συμβολικό και μόνο. Μετά, όσον αφορά τι δοκιμέ αναπτυσσόμενε χώρε, καλή ιδέα ότι αν ένα χορηγό θέλει να χρησιμοποιεί στοιχεία από δοκιμή που έγινε εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τότε η δοκιμή θα πρέπει να, να πληρεί τι προδιαγραφέ ε, που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, παρόλο που αυτό θα πρέπει να επεκταθεί ε, και σε διεθνεί ε, προδιαγραφέ που υπάρχουν όσο αφορά διδολογικά θέματα. Καλή είναι και η διάταξη για επιθεωρήσει από πλευρά των χωρών, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών και μια από τι καλύτερε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να την προσφυστεί στα ναρά το Κοινοβούλιο είναι και εξή. Το σύστημα εθνικής αποζημίωση. Γιατί? Διότι το το, το κόστος των ασφαλίσεων για κάποιες δοκιμές είναι σε αστυνομικά επίπεδα και ίσως έτσι να είναι απαγορευτικές διάφορες δοκιμές σε πανεπιστημιακό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά σπάνιες ασθένειες. Πολλά από τα δημόσια χρήματα ε, στις έρευνες χρησιμοποιούνται για ασφαλιστικά τέλη. Το κόστος της ασφαλείας είναι δυσανάλογο σε σχέση με τις αξιώσει. αξιώσεις. Το το, το, κόστος, ε, το τρέχον κόστος ε, θα είναι πολύ ψηλό, ε, θα μπορούσε να μειωθεί. Και υπάρχουν κάποιες χώρες που το εφαρμόζουν καλά, Δανία και άλλες χώρες και μπορούμε αυτές τις χώρες να χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα. Μετά, τι θέλω να αλλάξει από όλα αυτά. Θα ήθελα να αλλάξω πρώτα απ' όλα τους ορισμούς. πολύ σύγχυση δημιουργήθηκε όσον αφορά τους διάφορους ορισμούς ε, των κλινικών μελετών και κλινικών ε, δοκιμών. Χρησιμοποιούνται εναλλακτικά αυτοί οι όροι σε διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και προδιαγραφές προτείνουν να αλλάξουν οι ορισμοί των κλινικών μελετών, του clinical study, και να γίνει ε, μελέτη που σχετίζεται με ιατρικά προϊόντα. Το σκεφτήκαμε πολύ ενδελεχώς και μετά από πολλή συζήτηση φαίνεται ότι είναι καλύτερη διέξοδος. Επίσης πρότεινα κάποιες αλλαγές όσον αφορά την σχετικότητα που έχουν οι δοκιμές. Πολλοί δοκιμές που διενεργούνται σε, επί ομάδων που αντιπροσωπεύουν εκείνους που τελικά χρησιμοποιήσουν το φάρμακο. Οι γυναίκες πολύ συχνά υποεκπροσωπούνται σε δοκιμές, αλλά λιγότερα στοιχεία υπάρχουν όσον αφορά το πώς επηρεάζουν τα φάρμακα συγκεκριμένες γυναίκες. Άλλες δοκιμές αφήνουν εκτός ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι ε, έχουν μεγαλύτερες υπόκειται σε μεγαλύτερες επιπλοκές. Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση του πληθυσμού των δοκιμών δεν δίνεται άδεια για δοκιμή. Δεν έχει νόημα να γίνονται δοκιμέ σε ανθρώπου που είναι κάτω των 40 ετών όταν ε, το φάρμακο χρησιμοποιείται περισσότερο ή σε ανθρώπου που είναι πάνω από 50 ετών. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Μετά σε κάτι πολύ πιο επίμαχο. Το θέμα τη Επιτροπή των Δεντρολογικών Επιτροπών. Ε, πολλά υπόθηκαν για το ότι παράληψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και τι εννοεί όσον αφορά Προσπαθώ να, να το αποφύγει αυτό το θέμα των διοντολογικών επιτροπών, διότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω μεν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να είναι πολύ περιοριστική. Θέλω δε όμω να είμαι σίγουρη ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο αυτέ οι επιτροπέ δοντολογικέ στην αδειοδότηση των δοκιμών και για την εγγύηση τη ασφαλεία των ασθενών. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στην έκθεσή μου που ασχολείται με αυτό το θέμα και στο πρώτο τμήμα και στο δεύτερο τμήμα. Επίσης προτείνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει μια πλατφόρμα για να μπορούν να συνεργάζονται οι λογικές επιτροπέ και να ανταλλάσσουν βέλτιστε πρακτικέ σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το ζήτησαν πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι θετικότατη λύση και προσέγγιση. Τέλο, και εκεί εστιάζεται η έκθεσή μου. Διαφάνεια των αποτελεσμάτων, όσον τα αποτελέσματα των δοκιμών. Η έλλειψη διαφάνεια των αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών μείωσε την εμπιστοσύνη του κοινού στα φάρμακα και στην ιατρική. Ανεξάρτητοι πανεπιστημιακοί πολύ συχνά δυσκολεύονται να βρουν τα στοιχεία που θέλουν για να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα και να κάνουν συστηματικέ αναθεωρήσει. Και ακόμα χειρότερο, αν επιτυχεί αποτελέσματα δοκιμών δεν δημοσιεύονται ή δεν διατίθεται καθόλου. Πρέπει να βλέπουμε τα αποτελέσματα δοκιμών. Είτε είναι επιτυχεί οι δοκιμέ, είτε είναι ανεπιτυχεί. Οι δοκιμέ μπορούν να διενεργούνται επανειλημμένα πριν να γίνει γνωστό ότι είναι αποτελεσματικέ οι δοκιμέ και επικίνδυνε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μεγάλα βήματα προόδου όσον αφορά τη διαφάνεια. Προτείνει δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με πληροφορίε όσον αφορά τι δοκιμέ, είτε είναι επιτυχή είτε είναι επιτυχή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα πρόοδου. Όμω, κατά την άποψή μου, μια απλή σύνοψη των αποτελεσμάτων από τον χορηγό δεν είναι αρκετό. Θα μπορούσε να αμεροληπτεί ή να παραπλανεί. Θα ήθελα οι χορηγοί να πρέπει να δημοσιεύονται ολόκληρη έκθεση με τι κλινικέ δοκιμέ και τι μελέτε. Υπάρχουν διεθνεί προδιαγραφέ για εκθέσει για κλινικέ μελέτε ε, που, είναι, που πλήρως περιγράφουν το πώ διενεργείται η δοκιμή και ποια είναι τα πορίσματα τη δοκιμή και τα αποτελέσματα. Πολλοί χορηγοί ήδη ετοιμάζουν αυτέ τι εκθέσεις και υποβάλλονται όταν ζητούν αδειοδότηση για εμπορία ε, συμπεριλαμβάνεται απλούστευση σύνοψη, αλλά και πληρέστερα αποτελέσματα μπορούν να αναλυθούν και να ελεγχθούν από ανεξάρτητου ερευνητέ. Είναι σαφέ ότι οι ασθενεί αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε δοκιμή για να βοηθήσουν προχειρημένα φάρμακα να δημιουργούνται και για αυτού και για άλλου που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, όχι για να βοηθήσουμε μια ιδιαίτερη φαρμακοβιομηχανία. Λοιπόν, χρειάζεται επιμερισμό των γνώσεων, μοίρασμα των γνώσεων που θα οδηγήσει σε εμπιστοσύνη για τα φάρμακα και θα επιταχύνει και την ανάπτυξη διαφόρων θεραπείων που θα θρώσουν ζωέ. Και δεν θα υπονομεύσει την προστασία των δεδομένων, διότι όλα τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών θα διατίθενται αλλά ανώνυμα λοιπόν, εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την φυστάμενη νομοθεσία την πρόσβαση στα έγγραφα και εάν η χορηγή δεν είναι αρκετά διαφανής τότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν ε, πρόστιμα. Έχω την πεποίθηση ότι η Επιτροπή θα συμφωνεί ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαφάνεια. Ελπίζω και προσβλέπω σε συζητήσεις σήμερα και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας και προσβλέπω στην υποστήριξή σας στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mrs. Wilmot. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε κύριε Wilmot. Σκιώδης εισηγητές, ο Φίλιπ Ζουβέν καταρχήν από το... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ την εισηγήτρια και για την ποιότητα Τη έκθεσής τη και φυσικά και επικροτώ και την πρόταση της Κομισιόν. Πρόκειται για ένα κανονισμό για λόγους ο οποίους δεν πρόκειται να αναλύσω γιατί ξέρουμε ποια τύχη είχε η οδηγία που προτάθηκε πριν από 10 χρόνια περίπου. Οι πρόθεσμίε έχουν γίνει πολύ πιο σφιχτές, ίσως υπερβολικά, μεταξύ των στόχων που πρέπει να είναι εφικτοί και που είναι και μια προϋπόθεση για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι κλινικές δοκιμασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο στόχος μας είναι να διευκολύνουμε το έργο των ερευνητών, είτε είναι ε, ακαδημαϊκού χαρακτήρα, είτε είναι από φαρμακευτικές εταιρείες. Έχει δίκιο η κυρία Βίλμοντ όταν λέει ότι εμείς πρέπει να επαναφέρουμε την έννοια της Επιτροπής Δεοντολογίας για πάρα πολλούς λόγους. Μπορούμε να συζητήσουμε για πολλή ώρα για όλους αυτούς τους στόχους αλλά συμφωνώ για την ανάγκη να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τα δεοντολογικά θέματα. Υπάρχουν ορισμένα σημεία για τα οποία, τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τα οποία νομίζω πρέπει να βρούμε μια σειρά από Πρώτα απ' όλα το θέμα της κατηγοριοποίησης των ασθενών. Εδώ και πολλά χρόνια οι ερευνητικοί κύκλοι έχουν τροποποιήσει την προσέγγιση λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κατηγοριοποίηση επί τη βάση του κινδύνου ο οποίος προστίθεται από την έρευνα. Αυτό εμφανίζεται στον κανονισμό, στο σχέδιο κανονισμού, γιατί μιλάει για ε, low intervention, χαμηλό επίπεδο παρέμβασης η Κομισιόν στην πρότασή της. Στην πράξη όμως υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία δεν είναι ικανοποιητικά για, αυτή την, για αυτό τον ορισμό. Η Κομισιόν λέει να έχουμε τις δύο κατηγορίες της χαμηλής παρέμβασης και της μη χαμηλής παρέμβασης. Ενώ όλα τα διεθνή κείμενα, όλες οι διεθνείς συμβάσεις ακολουθούν μια άλλη κατηγοριοποίηση. Είναι κάπως τεχνικά αυτά τα πράγματα, υπάρχει μια τριπλή διάκριση. Καταρχήν, οι τεχνικές δοκιμασίες που αφορούν μονάχα τα φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν άδεια κυκλοφορία στην αγορά και που χρησιμοποιούνται μέσα στα πλαίσια της έγκρισής τους. Εδώ δεν υπάρχει καμία καινοτομία, απλώς γίνεται δοκιμασία των κλινικών πρακτικών. Η κατηγορία αυτή είναι μια κατηγορία πολύ χαμηλού κινδύνου που προκύπτει από την έρευνα. Εκεί υπάρχουν πολλές εθνικές διατάξεις που δεν ζητούν καμία πρόσθετη έγκριση παρά μόνο από την ε, Επιτροπή του. και δεν υπάρχει και η ανάγκη πρώτερη έγκριση από τι εθνικέ αρχέ. <clears throat> Ίσως λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια κατηγοριοποίηση, γιατί στι ε, έρευνες πολύ χαμηλή παρέμβαση για φάρμακα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και συγκρίνεται με ένα άλλο φάρμακο το οποίο βρίσκεται ήδη στην αγορά, δεν υπάρχει προστιθέμενος κίνδυνο και δεν υπάρχει λόγο να περιπλέξουμε την κατάσταση. Η Κομισιό λοιπόν προχωρά προ την κατεύθυνση αυτή των ε, κλινικών μελετών και δοκιμασιών χαμηλής έντασης. Χρησιμοποιεί όμως μια κατηγοριοποίηση που δεν συνάδει με τη διεθνή κατηγοριοποίηση και επίσης δεν αντλεί συμπεράσματα. Αν δείτε τον κανονισμό, το γεγονός ότι μια μορφή δοκιμών είναι χαμηλής παρεμβατικότητα, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα από το οποίο έλκεται από εκεί παρά, το, μόνο το γεγονός ότι ίσως είναι πιο μικρές χρονικές προθεσμίες. Ενώ μία από τις απόρριες θα μπορούσε να είναι η μείωση του επίπεδου απαιτητικότητας για τις εγκρίσεις, αλλά και επίσης για την ετικετοθεσία, αν χρησιμοποιείτε φάρμακα τα οποία βρίσκονται ήδη στο κοντινότερο σας φαρμακείο, δεν χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη ετικετοθεσία, επειδή χρησιμοποιούνται για μια κλινική μελέτη που δεν οδηγούν σε κίνδυνο για τον ασθενή. Η κατηγοριοποίηση λοιπόν είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης έχουμε τις ε, ε, μελέτες του άρθρου 31 που είναι αυτές σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δυστυχώς η σημερινή διατύπωση αυτού του άρθρου δημιουργεί προβλήματα γιατί δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα ουσιαστικά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Λέει το άρθρο 31 ότι η έρευνα αυτή μπορεί να γίνει σε κατεπίγουσες περιπτώσεις το άρθρο 32 όχι 31 μόνο αν δεν υπάρχει κανείς ε, νομικός εκπρόσωπος. Αυτό σε πάρα πολλέ περιπτώσει κάνει απόλυτα δύνατη να γίνει η έρευνα. Α υποθέσουμε ότι εδώ σε αυτή την αίθουσα πέφτει ξερό κάποιο και παθαίνει καρδιακή προσβολή. Η ανάληψή του πρέπει να γίνει στα επόμενα δευτερόλεπτα. Κάθε δευτερόλεπτο που χάνεται δημιουργεί πρόβλημα. Αν αποφασίσετε να κάνετε μια κλινική έρευνα για να δοκιμάσετε μια νέα μέθοδο καρδιακού μασάζ, τότε βάσει του άρθρου 32 δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της οικογένειας, κάποιος ε, νόμιμος εκπρόσωπος. Πρέπει να τροποποιήσουμε λοιπόν το κείμενο ώστε να μπορεί κανείς να κάνει μια τέτοια έρευνα και στη συνέχεια να ζητήσει την ε, έγκριση του εκπροσώπου γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος για να ζητήσει κανείς την έγκριση. Η έγκριση αυτή μπορεί να απαιτήσει ένα τέταρτο, μισή ώρα, μπορεί και περισσότερο. Επίσης, το εδάφιο 1ε του άρθρου 32 λέει ότι οι κλινικέ αυτέ μελέτε θα πρέπει να οδηγούν σε ένα ελάχιστο κίνδυνο. Δεν ξέρω τι είναι ελάχιστο κίνδυνο. Υπάρχει το λεγόμενο το εγκεφαλικό έμφραγμα, μια μορφή δηλαδή συμφόρηση, η οποία για πολύ καιρό δεν είχαν κανένα φάρμακο για την αντιμετώπιση του. Τώρα υπάρχουν φάρμακα που ανοίγουν τις αρτηρίες και οξυγονώνεται και πάλι ο εγκέφαλο. Αυτό βέβαια έγινε με κλινικές μελάτε που ήταν επικίνδυνες γιατί 10% των ασθενών οδηγήθηκαν σε εγκεφαλικές αιμορραγίες. Τα άλλα 90% των ασθενών επωφελήθηκαν από αυτό το φάρμακο. Αυτό το φάρμακο τώρα έχει εγκριθεί να κυκλοφορήσει. Αν λέτε λοιπόν ότι ο κίνδυνος πρέπει να είναι ελάχιστο, τέτοιου είδου έρευνε είναι αδύνατε. Ο κίνδυνο θα πρέπει να είναι ανάλογο με το προσδεκόμενο όφελο. Μακρηγόρησα κύριε Πρόεδρε, Κάτι ακόμα για την έκθεση της κυρίας Βίλμοτ. Πρέπει πράγματι να υπάρχει και μια πλήρης έκθεση στη διάθεση του κοινού. Το θέμα όμως της πληρότητος είναι ένα πρόβλημα. Κυρία Βίλμοτ λέτε κάτι το οποίο έχει τεχνικό χαρακτήρα, <clears throat> να λέτε, να λέτε ότι η έκθεση πρέπει να είναι τόσο πλήρης που να αντανακλά τα πρότυπα τα οποία αναφέρονται, τα σε αστρία κτλ. Αυτό μπορεί να είναι πράγματι πλήρες, αλλά αυτό θα οδηγήσει σε προβλήματα για τους ακαδημαϊκούς που κάνουν αυτές τις μελέτες. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια εκθέση πιο πλήρη από αυτή που θέλει η Κομισιόν, αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που να δημιουργεί προβλήματα στου ερευνητέ. Αντίθετα, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι παράλληλα να πούμε, όπω είπατε, ότι όλα τα στοιχεία θα πρέπει να είναι στη διάθεση όλων αυτών που θέλει να τα επανεξετάσει. Όταν λέμε ότι τα δεδομένα θα πρέπει να είναι πλήρω στη διάθεση του κοινού, Πρέπει να ξέρετε ότι σε μία έρευνα όλα τα δεδομένα σημαίνει χιλιάδες και χιλιάδες σελίδες. Το να δώσουμε τώρα στο κοινό αυτές τις σελίδες δεν βοηθάει στην κατανόηση και δεν κάνει πιο διάφορα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζούδα. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τους άλλους ομιλητές να είναι κάπως σύντομοι, αλλιώς ε, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αντωνία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Κλένης για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης που αντιμετωπίζει τα βασικότερα ζητήματα του σχεδίου κανονισμού. Εμείς χαιρετίζουμε την πρόταση και τη γενική της αρχιτεκτονική που προέκυψε μετά από εκτεταμένη διαβούλευση και η οποία κατά την απόψή μου είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για τους ε, στόχους που έχουμε. Όσον αφορά το σχέδιο έκθεσης, καλωσορίζω ιδιαίτερα τις αλλαγές που έχουν εισαχθεί στα εξή σημεία. Τα προσόντα και τον ρόλο των Επιτροπών Ηθικής, ε, η διαβούλευση, το ότι πρέπει να ενημερώνουν οι να λαμβάνεται υπόψη η υγεία και η ευημερία τους, ε, οι όροι που προστίθενται στις κλινικές δοκιμές, ειδικά για τα καινοτόμα φάρμακα. Επίσης ε, στηρίζουμε την αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν για το χρονοδιάγραμμα έγκρισης, το Εθνικό ε, Σύστημα Αποζημίωσης και τις προβλέψεις που υπάρχουν για δοκιμές σε τρίτες χώρες. Θα αναφερθώ τώρα στα βασικά σημεία που μας απασχολούν για να καταλήξουμε σε μια βέλτιστη θέση του Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα για τις επιτροπές ηθικής, όπως ήδη αναφέρθηκε, στηρίζω τις ε, διευκρινήσεις που προτείνει η συγγήτρια για να διασφαλιστούν όσοι λένε πως οι επιτροπές αυτές ε, ε, είχαν ξεχαστεί από την Κομισιόν. Δεν ισχύει αυτό και υποστηρίζουμε επίσης την χωριστή ψηφοφορία. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο η αρχή πως καμία κλινική δοκιμή δεν πρέπει να ξεκινήσει σε μια χώρα χωρίς την ε, έγκριση μιας εθνικής ηθικής επιτροπής πρέπει να διατηρηθεί, αλλά βεβαίως ε, είναι και ένα ζήτημα επικουρικότητας, δηλαδή μια απόφαση μια τέτοια επιτροπή δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ε, διαδικασία σε άλλο κράτο μέλο. Η συζήτηση νομίζω λοιπόν αυτή θα πρέπει να ε, ηρεμήσει λίγο και να εμπιστευτούμε το επίπεδο των επιτροπών σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζω την πρόταση της Γκλένης για την στήριξη του έργου των επιτροπών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών παρόλα αυτά. εάν εγκριθεί ένα φαρμακευτικό προϊόν, θα μπορέσει να ασχοληθεί σε ολόκληρη την Ένωση ανεξαρτήτως του που έχουν γίνει οι δοκιμές. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όσον αφορά λοιπόν τη διαφάνεια και την διαθεσιμότητα των δεδομένων, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και καλωσορίζω την πρόταση παρά το ότι θα ήθελα κάποιε περισσότερε διευκρινήσει για το τι εννοούμε όταν λέμε ε, έκθεση κλινική μελέτη και ποιε πληροφορίε θα είναι διαθέσιμε σε ποιον. Επίσης, πρέπει να θέσουμε τρία ερωτήματα. ποιο είναι ο στόχο μας όσον αφορά την διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, τι μπορεί να αποκαλυφθεί πριν και μετά την ε, ε, έγκριση της ε, εμπορίας και ποιες πληροφορίες είναι χρήσιμες και σε ποιον. Μετά από αυτά τα ερωτήματα λοιπόν δεν θεωρώ πως το να δώσουμε στο κοινό ακατέργαστα δεδομένα στο διαδίκτυο. Δεν νομίζω πως θα χρησιμεύσει τίποτα όμως. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να έχουν κάποια σημασία από τη μακροπρόθεσμη σκοπιά της δημόσιας υγείας, οπότε θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για στόχους έρευνας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τις πληροφορίες ε, που δίνονται πριν δοθεί η άδεια εμπορίας για να μην έχουμε ε, πρακτικές ε, του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και η διαχείριση των πληροφοριών που θα διατεθούν και εδώ πέρα καλωσορίζω τις απόψεις Κομισιόν τέλος. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων ε, την οποία θα εξετάσουμε Ένα άλλο ζήτημα θα ήθελα να αναφέρω. η συμβατότητα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο φαρμακοεπαγρύπνησης, η αποτελεσματικότητα των ελέγχων μετά την αδειοδότηση και βεβαίως τα γενώσιμα φάρμακα και τα πειράματα που γίνονται σε ε, υγιείς σας ευχαριστώ. Η κυρία Όκον από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Βίλμοτ για τη θαυμάσια εργασία της. Είναι πολύ καλή βάση για την περαιτέρω εργασία μας. Να υπογραμμίσω τώρα το εξής. Πρωτού πω οτιδήποτε άλλο. ότι οι κλινικές μελέτες είτε είναι επιτυχής είτε όχι, δίνουν αποτελέσματα που δεν ανήκουν στους επιστήμονες, αλλά στην ανθρωπότητα, όχι στις εταιρείε, όχι στους ερευνητές. Γιατί έχουν βάλει την υγεία τους και τα σώματά τους στον τορβά οι εμπλεκόμενοι στις κλινικές μελέτες. Επομένως, από δεοντολογική άποψη δεν είναι ηθικό να κοιτάζουμε μονάχα τα οικονομικά συμφέροντα και όχι τη δεοντολογία και την ηθική. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να διατρέχει όλες τις προσεγγίσεις μας σε αυτά τα θέματα. Ο κανονισμός αυτός είναι μια ιστορική ευκαιρία για να μπορέσουμε να τονίσουμε αυτό το γεγονός. Μια φορά και για πάντα. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια τα οποία μπορούν να εξοικονομηθούν αν υπάρξει σωστή ρύθμιση με αυτόν τον κανονισμό και μπορούμε να σώσουμε και χιλιάδες ζωές με ένα σωστό κανονισμό. Εγώ ήμουν πρόσφατα στην, στο Λονδίνο στην υπηρεσία εξέταση των φαρμακευτικών σκευασμάτων, στην EMA μαζί με την Επιτροπή μας και από ό,τι καταλαβαίνω αυτή είναι και η δική τους θέση. Δεν ενδιαφέρονται στο να υπάρχει, να υπάρχει εμπιστευτικότητα για τα αποτελέσματά τους και δεν τους ενδιαφέρει <clears throat> οποιοδήποτε άλλο συμφέρον παρά μόνο το συμφέρον της ανθρώπινης υγείας και το κοινό συμφέρον. Είναι σκανδαλώδες το ότι υπήρξε μήνυση κατά τη CMA e από φαρμακευτικές εταιρείες για την διάδοση των αποτελεσμάτων. Είναι σκάνδαλο, δεν μπορώ να πω τίποτα λιγότερο από όλα αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θέλει η φαρμακευτική βιομηχανία να υποστηρίξει την πλήρη αποκάλυψη των αποτελεσμάτων. Αν υποστηρίζουν τη διαφάνεια, ακόμα καλύτερο. Αυτοί όμως οι οποίοι θέλουν πράγματι να συμπεριφέρονται με σωστό τρόπο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τον ίδιο συνθήκων ανταγωνισμού με τους υπόλοιπους. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυτή τη διαφάνεια που πρεσβεύουν οι ίδιοι. Και όπως έχετε κατανοήσει πλέον, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η απόλυτη διαφάνεια ακόμα και σε ό,τι αφορά τα ακατέργαστα δεδομένα. Πολλοί έχουν εκφράσει ανησυχίες σε σχέση με τον τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα δεδομένα. Αν έχουμε αυτά τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή και υπάρχει δημόσια πρόσβαση σε αυτά τα γεγονότα, Αυτό δεν είναι αρνητικό. Ναι, πρέπει πράγματι όλοι να έχουν πρόσβαση σε όλα τα ακατέργαστα στοιχεία. Ένας δημοσιογράφος της Guardian κοίταξε πώς γίνονται αυτές οι κλινικές μελέτες και ανακάλυψε ότι γιατί τα αντικαταθλιπτικά μπορούν να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα... στους εφήβους. Αυτό είχε μείνει μυστικό. Γιατί λέγανε ότι αυτά τα φάρμακα βοηθούν τους ε, νέους, τους teenager. Αντίθετα ήταν επικίνδυνα και πολλά πολλά παιδιά έχασαν, πολλοί νέοι έχασαν τη ζωή τους λόγω αυτών των φαρμάκων. Ένας δημοσιογράφος λοιπόν τα βρήκε όλα αυτά. Αν εμείς σαν πολιτικοί φοβόμαστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δεν αξίζουμε τίποτα. Πρέπει να πούμε λοιπόν στη φαρμακευτική βιομηχανία ότι εάν συμπεριφερθούν σωστά, τότε μπορούν να αντέξουν ακόμα και τους κακούς δημοσιογράφους και εδώ είχαμε ένα πολύ κακό δημοσιογράφο. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους ερευνητέ, θέλουμε να υποστηρίξουμε την ηθική βιομηχανία και πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα όντα. Αυτά λοιπόν ήθελα να αναφέρω υπό σχολείων. Ελέγχθηκαν πολλά για τις επιτροπές δεοντολογίας που είπαν ότι στη Γερμανία η Bundestag έχει εγκρίνει μια στεναρή νομοθεσία για τις επιτροπές δεοντολογίας στα κρατήρια της Γερμανίας και αυτό θα πρέπει να μας χαροποιήσει. Και πρέπει να επικροτήσουμε αυτά τα οποία λέει η Γκλέλης Φίλμοντ στην έκθεσή της. Δεν θέλω να προσθέσω και άλλα ερωτήματα σε αυτά τα οποία υπάρχουν. Απλώς ελπίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε την εστίασή μας στους ανθρώπους. Περί αυτών πρόκειται. Έχουμε πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς υγείας και αυτό είναι θέμα που αφορά τους ανθρώπους γιατί αν δαπανούμε πολλά χρήματα σε φάρμακα που είναι άχρηστα όπως το ταμιφλού, έχουμε λιγότερα χρήματα για τα φάρμακα που πράγματι χρειαζόμαστε. Είναι λοιπόν και αυτό ένα θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ο κ. Τσάβερνόχα από του Ευρωπαίου Συντελικού δεν είναι εδώ πέρα. Αλλά βεβαίω ε, τον αντικαθιστά η συνάδελφό του. Α, ε, μια που ξεκινήσαμε με τα Δανέζικα, λέει η κυρία Ρόσμπαχ, να συνεχίσω κι εγώ. Δυστυχώ ο αδελφό μου βεβαίω ε, δεν είναι εδώ πέρα σήμερα, αλλά στηρίζει ε, 100% την πρόταση του εισηγητή. Αλλά οπωσδήποτε θα προτείνουμε κάποιες ε, τροπολογίες. Αλλά ο συνάδελφος οπωσδήποτε στηρίζει τον εισηγητή. Θέλω να πω τώρα στη Μαργαρίτα πως σε ευχαριστούμε. Δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά αυτή τη φορά συμφωνούμε. Και ελπίζουμε όσοι ε, είναι στη φαρμακευτική βιομηχανία να μην αρρωστήσουν ποτέ γιατί θα είναι στην ίδια κατάσταση με εμά. Και θα χρειάζονται προϊόντα που δεν λειτουργούν ίσως ή ε, έχουν πάρει μια λάθος τροπή. Ε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μας απασχολούν, το κρέας των αλόγων ε, και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος θεωρεί πως πρέπει να κάνει τέτοιες δραστηριότητες μόνο και μόνο για να οικονομήσει. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρόσμπαχ. Η κυρία Σούσαλ, εκ μέρους της ΚΟΥΕ, είναι η επόμενη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είναι ένα τόσο πολύπλοκο θέμα και τόσο αχανές, αλλά τόσο σημαντικό και εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πτυχές αυτού του θέματος, την πτυχή της ηθικής και της ιδεοντολογίας και επίσης την πτυχή της διαφάνειας. Εγώ πιστεύω, όπως και η ομάδα μου, ότι η πρόταση της Κομισιόν με την αρχική της μορφή που συζητούμε εδώ είναι μια υποχώρηση ή μια υπαναχώρηση σε σχέση με τις αρχές που πρέπει να διέπουν την ιατρική έρευνα. δεν είναι δική μου αυτή η διαπίστωση. Η Παγκόσμια Ιατρική Οργάνωση στην γρομοδότηση που έστειλε για αυτήν την ε, πρόταση και που πήρα και εγώ όπως όλοι οι συνάδελφοι και δεν έφτασε μόνο σε αυτή η γνωμοδότηση λέει το εξής η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη τις βασικές ειδικές αρχές που βρίσκονται στην δήλωση του Ελσίνκη. Η πρόταση αυτή της Κομισιόν δεν έχει σαφήνεια σε σχέση με την ανάγκη να υπάρξει έγκριση των κλινικών μελετών από ανεξάρτητες επιτροπές δεοντολογίας. Δεν υπάρχει στην πρόταση λοιπόν αυτή η ανάγκη πρώτερης έγκρισης και επίσης υπάρχει ένας άλλος φορέας που είναι πολύ σημαντικός, η ΙΟΡΕΚ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των ε, Ηθικών Διοντολογικών Επιτροπών για την Έρευνα, λέει τα ίδια πράγματα περίπου. Λέει ότι η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να εμπλέκονται οι Επιτροπές Δεοντολογίας και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν και διάφορες πτυχές που συνδέονται με αυτό το σημείο συγκεκριμένα. Η δυνατότητα να υπάρξουν διαφωνίες ή αυτοεξαίρεσης από τα κράτη-μέλη είναι πολύ περιορισμένες και δεν λαμβάνονται υπόψη ηθικές πτυχές των κλινικών μελετών εδώ. Φοβάμαι λοιπόν ότι με όλα αυτά δημιουργείται ένας κίνδυνος αυτοί οι οποίοι χορηγούν και χρηματοδοτούν τις κλινικές μελέτες να ψάχνουν χώρες οι οποίες έχουν λιγότερο υψηλές προδιαγραφές για να κάνουν και τις κλινικές τους μελέτες. Και όπως προτείνεται από την Κομισιόν, η έγκριση ενός κράτους μέλους ισχύει και για τα άλλα κράτη-μέλη για να γίνει η μελέτη. Επίσης, η δυνατότητα τα κράτη να ελέγχουν τις ε, προτάσεις για μελέτες είναι πάρα πολύ στενά τα χρονικά όρια και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και δημιουργεί και κίνδυνο για την σωστή εφαρμογή των πρωτοκόλων των μελετών. Το θέμα της έγκρισης, της έγκρισης εν γνώση και εγγράφος είναι πολύ σημαντικό. Κατανοώ ότι υπάρχουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αλλά σε μια φυσιολογική κλινική μελέτη είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει μια εμπεριστατωμένη έγκριση από τους ενδιαφερόμενους. Και αυτό δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι προηγουμένω, για τα θέματα της διαφάνειας και την ανάγκη να υπάρχει πρόσβαση όλων στα αποτελέσματα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Είναι φανερό ότι για τα δεδομένα των ε, κλινικών μελετών θα πρέπει να υπάρχει φυσικά όλη η απαραίτητη προφύλαξη για την μη αποκάλυψη προσωπικών γεγονότων. Θα πρέπει να είναι ανωνυμοποιημένα όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το κοινό και οι άλλοι ερευνητέ να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα, τα λεπτομεριακά αποτελέσματα των ερευνών και όχι μονάχα σε συνοπτικά αποτελέσματα όπω γίνεται συνήθω στι κλινικέ μελέτε. η πρόταση της η Κομισιόν λέει ότι οι κλινικές μελέτες έχουν μειωθεί σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έγκριση της οδηγίας. Αλλά στην πρότασή της δεν αναφέρει πουθενά κάποιο επιστημονικό άρθρο το οποίο επικυρώνει και επιβεβαιώνει τα στοιχεία τα οποία παραθέτει η Κομισιόν. Θα ήθελα η Κομισιόν να μας δώσει και τα στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν αυτή τη μείωση των ε, κλινικών μελετών, εάν τα έχει στη διάθεσή της. Αλλά ακόμα και αν έχει δίκιο η Κομισιόν, πιστεύω ότι δεν πιστεύω ότι με το να μειώσουμε τις δεοντολογικές απαιτήσεις από τις κλινικές μελέτες που θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των μελετών και θα προωθήσουμε την εφαρμογή αυτών των μελετών. Αυτό δεν είναι ηθικό, δεν είναι λογικό, δεν είναι ανθρώπινο να θεωρούμε ότι με το να παίζουμε με τις δεοντολογικές απαιτήσεις θα μπορέσουμε να προωθήσουμε περισσότερες μελέτες. Επίσης θα ήθελα να πω στην εισηγήτρια θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία βέβαια η έκθεσή της για ορισμένα τμήματα της έκθεσης της συμφωνώ, για όλα όχι βέβαια. Θα παρουσιάσει η ομάδα μας κάποιες τροπολογίες, όχι μόνο για τα θέματα τα οποία έφεραν και για άλλες. Και είμαστε πάντα στη διάθεση της για να συνεργαστούμε με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και με την ίδια φυσικά για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την πρόταση κανονισμού μια καλή πρόταση η οποία προασπίζεται τα συμφέροντα των ατόμων και προασπίζει και τις ηθικές πτυχές της, ε, των κλινικών μελετών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπερέχουν τα οικονομικά συμφέροντα της ανάγκης θεοντολογίας στις ε, ηθικές, στις ε, κλινικές μελέτες και σας λέω και πάλι με έτοιμη να συνεργαστώ για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πρόταση που ευράζεται ε, σε αυτές τις ηθικές αρχές. Και σας υπενθυμίζω τη γνωμοδότηση σχετικά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ιατρών. Ευχαριστώ. πολύ κυρία Σούσα. Πάμε στους τελευταίους 7 ομιλητές. Έχουμε 40 λεπτά που μας απομένει αυτό το θέμα και τα τρία αναπομένοντα σημεία. Δύο λεπτά λοιπόν ο καθένας. Ο Πέτερ Λίζε ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι ε, πρέπει να ξαναπώ πως ο χρονικός περιορισμός πρέπει να τίθεται στην αρχή και όχι στη μέση της συνεδρίασης. Χαίρομαι για το είναι η κυρία Γουλμότ και ο Φιλίπ Ζουβέν οι αρμόδιοι για το θέμα αυτό και ο συγητές και υπάρχουν πάρα πολλά μονομερή δημοσιεύματα. Ε, χτες ε, αναφερθήκατε, αναφέρθηκε μία συνάδελφο σε αρνητική κριτική στα ΜΜΕ της Γερμανίας ε, για την πρόταση Κομισιόν. Ε, και ενώ υπάρχουν πάρα πολλά θετικά σημεία στην πρόταση της Κομισιόν. αλλά έτσι όπως έχει ε, κάνει την πρόταση Κομισιόν δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Χρειαζόμαστε επιγόντως αλλαγές. Και εγώ δεν θα υπερψηφίσω εάν δεν δούμε επιγόντως την προστασία των ατόμων τα οποία δεν μπορούν από μόνα τους να κρίνουν και να αποφασίσουν. Το είχαμε διαπραγματευτεί το 2000. Αρχικά το Κοινοβούλιο είχε πει στην πρώτη ανάγνωση πως θα πρέπει ε, για παιδιά και πνευματικά ε, καθυστερημένους, να μην γίνονται σε παιδιά και πνευματικά καθυστερημένους, να μην γίνεται καμία κλινική δοκιμή και η Κομισιόν το χαλάρωσε. Δεν είναι δυνατόν να χαλαρώνουν οι κανόνες για τα παιδιά. Τι είπα να πει, τους το ζήτησαν. Και άλλοι ζήτησαν άλλα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε στην κατάσταση του 2001. Ε, για τις Εθνικές Επιτροπές στηρίζω την κυρία Παρβάνοβα, πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και η διαδικασία για το πώς συνεργάζεται το κράτος που έχει την ηγεσία με τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, το ένα κράτος μπορεί να πει ναι, τα υπόλοιπα τέσσερα να πούνε όχι και παρόλα αυτά επειδή ένα κράτος έχει τον ηγετικό ρόλο η απάντηση να είναι ναι. Ε, δεν είναι διαδικασία αυτή και έχω μία παράκληση να ξαναδούμε το χρονοδιάγραμμα. Το θέμα είναι περίπλοκο και μπορεί να μην είναι όλοι οι κριτικοί δικαιολογημένοι, αλλά θα έχουμε μεγάλη πίεση. Αυτό θα ήθελα να έχουμε χρόνο για να διατυπώσουμε τις τροπολογίες και να τις συζητήσουμε κιόλας. Ευχαριστώ. Κρίστελ Σχαλντεμόζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και θα μιλήσω για λιγότερο από δύο λεπτά. Ξεκινώντα, θα ήθελα να πω στην Κλένη Βίλμοτ ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η έκθεση. Είναι ισορροπημένη, εξισορροπεί την προστασία των ασθενών με τις αποτελεσματικότερες κλινικές δοκιμές. Ο λόγος που παίρνω το λόγο είναι για να υποστηρίξω κάποιους συναδέλφους που είπαν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά ε, τις κλινικές δοκιμές. Νομίζω ότι η υποβολή ε, εκθέσεων για τις δοκιμές, αυτή η πρόταση είναι καλή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε περισσότερο το ότι πρέπει να δίνουμε πρόσβαση όχι μόνο στην έκθεση που αφορά τις δοκιμές, αλλά και τα δεδομένα τα ίδια. Το ξέρω ότι μπορεί να συζητηθεί το θέμα των εμπορικών συμφερόντων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ανεξάρτητοι ερευνητέ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη, στο υλικό, στα δεδομένα. Πρέπει να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι οι πολίτες και οι ασθενείς έχουν δικαίωμα στη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Νομίζω ότι είναι καλή έκθεση και ελπίζω να πετύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία των ασθενών. Η Κορίν Λεπάζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν να αποκατασταθεί η Επιτροπή Διοντολογία. Οι Επιτροπές Διοντολογία είναι απαραίτητο αυτό. Οι προθεσμίες είναι πάρα πολύ σύντομε διότι οι απόφαση θα πρέπει να λαμβάνονται χωρίς τα κράτη-μέλη να μπορούν να αποφανθούν. Αν είναι αποδεκτό, αν υπάρχει έγκριση των δοκιμών από την Ιντολογική Επιτροπή. Ε, ε, αυτό είναι δεκτό, το άλλο δεν είναι δεκτό. Κάτι άλλο που δεν αναφέρθηκε είναι το ποπενός ορισμός εκείνου που δεν αναφέρεται εκείνο που δίνει τα χρήματα. Οι εταιρείε που αναθέτουν υπεργολαβία για τις έρευνες σε διάφορες εταιρείε απαλλάσσονται από τις ευθύνε. Νομίζω ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα να έτσι ισχύει. Τρίτον, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες έτσι μας είπε η κυρία Άουκεν, είναι απαραίτητο να καθορίσουμε τον πρώιμο εντοπισμό αρνητικών συνεπιών Έχουμε αρκετά προβλήματα στην Ευρώπη και πρέπει να το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα και τέλος να αποθαρρυνθώ η παραγωγή μη δεοντολογικών ε, προϊόντων σε τρίτες ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ελπίζω ότι παρέμεινα στα όρια το χρονικά. Ευχαριστώ κύριε Λεπάς. Η Φρανσουάς ε, Γκροστέτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι πρόκειται περί κανονισμού ε, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία που είχαμε γιατί ήταν καταστροφικά τα αποτελέσματά της και είδαμε σημαντική υποχώρηση, μείωση των κλινικών δοκιμών στην Ευρώπη και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε δύο τμήματα. Ένα τμήμα αφορούσε τις τεχνικές και επιστημονικές τυχές και το άλλο τμήμα αφορούσε τα ηθικά θέματα και αυτό άπτεται της επικουρικότητας. Δεν πρέπει να κολλήσουμε στο θέμα των επιτροπών των διδολογικών. Λέμε ναι λοιπόν για τη δεντολογία, όμως θα λάβουμε υπόψη και το πνεύμα του κειμένου. Όσον αφορά την αναλογική προσέγγιση των κίνδυνων που εισάγεται στην πρώτη κανονισμού, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι καλό. Έχουμε μια κατηγορία δοκιμών μικρής παρέμβασης που μπορεί να μειώσει το διοικητικό άχθος για τις μελέτες χαμηλού κινδύνου και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Επανειλημμένα η πρόταση κανονισμού προβλέπει ότι η λήψη απαντήσεω από πλευρά των διαφόρων αρχών αυτό θεωρείται ότι είναι θετική ανταπόκριση, δηλαδή θεωρείται σιωπηρή έγκριση, σιωπηλή συνένεση και είναι ένα μηχανισμό εκτός για την πρόσβαση στα δεδομένα. βεβαίω χρειάζεται διαφάνεια, διαφάνεια που σέβεται όμω, τα συμφέροντα τη έρευνα, δηλαδή οι δημοσιοποιημένε πληροφορίε θα πρέπει να στατεύουν τα εμπιστευτικά χαρακτήρα, τα προσωπικά και εμπορικά δεδομένα. Να αποφευθεί η στιγματοποίηση, στιγματισμό των ασθενών που συμμετέχουν στι κλινικέ ε, δοκιμέ και να μην υπάρχει θέμητο ανταγωνισμό. Είναι κάτι επαχθέ, η έρευνα δαπανηρό και θα πρέπει να διαφυλάσσεται η πνευματική διοκτησία. Σε περίπτωση σπάνια ασθενεία και υπερβολικά σπάνια ασθενεία, η δυσκολία κλινικών δοκιμών πολύ συχνά συνδέεται με το μικρό αριθμό ασθενών για κάθε ασθένεια. Άρα και υπάρχει και γεωγραφική κατάτμιση και διασκορπισμός. Θα πρέπει να βάλετε υπόψη και η διάδοση, πόσο διαδομένη μια ασθένεια, να βάλετε υπόψη στο κείμενο για να δείτε προτεραιότητα σε κάποιε δοκιμέ κλινικέ από κράτη-μέλη. Κυρίω για τι σπάνιε και πάρα πολύ σπάνιε ασθένειε. Αναφερθήκαμε στην παιδιατρική. Στην παιδιατρική υπάρχουν καρκίνοι υπερβολικά σπάνιοι που πλήττουν τα πολύ μικρά παιδιά και θα πρέπει σε αυτέ τι περιπτώσει να υπάρχουν κλινικέ δοκιμέ, να προβλέπονται κλινικέ δοκιμέ χωρί να είναι πολύ περιορισμένοι οι όροι κάτω του οποίου θα δεξάγονται. Ευχαριστώ κύριε Γκοστέτ. Κάρο Σλούτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση κυρία Γουίλμοντ πήγαινε στη σωστή κατεύθυνση και άλλο θέλω όμω και άλλο, περισσότερα. Σήμερα έχουμε πολλέ αστοχίες, υπάρχουν πολλά αρνητικά αποτελέσματα τα δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ, οπότε είναι απαραίτητη η διαφάνεια. Επίσης όμως και μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Όταν λέει κανείς ποια είναι τα βασικά αποτελέσματα, αυτό θα πρέπει να παραμείνει το βασικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Αν θέλετε να μετρήσετε τον, τη μείωση των ε, καρδιακών προσβολών, δεν μπορείτε να αλλάξετε στον δρόμο και να πείτε ότι μετράτε τη χοληστερίνη στο αίμα. Το ίδιο και με τις υποομάδες. Θα πρέπει να πει κανείς στην αρχή ποιε είναι οι ομάδες στόχου. Δεν μπορεί μετά να διαλέγει κανείς τα στοιχεία τα οποία από στατιστικές συγκυρίες και συμπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Πρέπει από την αρχή να αναφέρετε ποιες είναι οι διάφορες ομάδες στις οποίες κατανέμετε τους ασθενείς, ώστε να μην μπορείτε να διαλέξετε στην αρχή αυτό που σας βολεύει. Πρέπει να έχουμε και κάποιες απαιτήσει για τις υπεργολαβίες και τις μελέτες που γίνονται σε τρίτες χώρες. Αν θέλετε έγκριση κάποιου φαρμακευτικού σκευάσματος στην Ευρώπη, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι κανόνες ανεξάρτητα από το πού γίνεται η έρευνα. Αν θέλετε να έχετε ένα χάπι το οποίο εγκρίνεται στην Ευρώπη θα πρέπει να δημοσιεύσετε και τις μελέτες άλλων σε ίδιες συνθήκες με την Ευρώπη. Αν κάνουμε λοιπόν αυτές τις αλλαγές όπως προτείνεται και με τις τροπολογίες που ελπίζω ότι θα εγκρίνουμε, ελπίζω μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο τρόπο προσέγγισης που βασίζεται περισσότερο στην επιστημονική γνώση στην Ευρώπη. Γιατί αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί κανείς στατιστικές συμπτώσεις για να προωθήσει ένα αποτέλεσμα. Και επίσης ε, όταν δεν εγκρίνεται κάποιο φάρμακο για, ένα, για το συγκεκριμένο σκοπό του, αλλά χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα και οι έρευνες για τις διάφορες ομάδες να δημοσιεύονται ακόμα και αν δεν είναι για τον κύριο σκοπό του φάρμακου αλλά μπορούν να έχουν αποτελέσματα θετικά για άλλους λόγους. Ο Ρίχαρτ Ζέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε πως η ασφάλεια είναι ο βασικός στόχος αυτής της οδηγίας και ειδικά για περιπτώσεις ασθενών που δεν μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους. Πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο πως θα πρέπει τα πειράματα να, να μειωθούν στο ελάχιστο και να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματά τους και για άλλες ε, περιπτώσεις. Και πρέπει εδώ πέρα να προωθήσουμε τη δυνατότητα της συνεργασίας και της χρήσης των διαφόρων μελετών στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό και για άλλους σκοπούς. Και με αποζημίωση βεβαίως, αλλά πρέπει να υπάρξει μία βάση δεδομένων ή ένα δίκτυο βάσεων δεδομένων και εδώ πέρα νομίζω πως η Κομισιόν πρέπει να παίξει τον ρόλο της για να δούμε πώς θα βελτιωθεί αυτό το σύστημα για να α, ε, μπορέσουμε όπως να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά ως το δυνατόν ευρύτερα. Επίσης σημαντικό είναι πως ε, συχνά τα νέα μέσα αυξάνονται με ρυθμό αλματώδη και αυτό βοηθάει στην διάθεση των νέων φαρμάκων. Επίσης ε, δεν είναι σωστό να γίνεται η έρευνα εκτός Ευρώπης και για ηθικούς αλλά και για επιστημονικούς λόγους. Ε, βεβαίως θα πρέπει παντού να τηρούνται οι ίδιες προδιαγραφές αλλά θεωρώ πως ε, είναι καλύτερες οι δυνατότητες ελέγχου εντός της Ευρώπης παρά εκτός ε, και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Επίσης σημαντικό είναι να λαμβάνουμε υπόψη και τον ασθενή, να του δίνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο είπε η Γκλένις Βίλμοτ για να επεκτείνουμε ακριβώ αυτή την πτυχή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ζέιμπερ. τελευταία ομιλητή, κυρία Χιούμπνερ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό, το θέμα των ε, κλινικών ε, δοκιμών. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να οδηγήσει σε πλήρη διαφάνεια. Πρέπει όμως να ακολουθούνται και συγκεκριμένες διαδικασίες για τις δοκιμές. Διότι αυτό το οποίο ε, αναφέρεται είναι η παθολογία. Εμείς όμως πρέπει να συζητήσουμε και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις κλινικές δοκιμές. Δοκιμές που διενεργούνται από εγκεκριμένου φορείς και ερευνητικά κέντρα και δεν διενεργούνται από εγκληματικές οργανώσεις, παραδείγματος χάρη. Το αλογίσιο κρέας δεν απαγορεύεται αλλά πρέπει να ενημερώνεται ο καταναλωτής για το τι τρώει. Δεν μπορούμε να λέμε ότι φταίνε για όλα οι φαρμακευτικές εταιρείες. Πρέπει να εστιαστούμε στον ασθενή, να δούμε τι γίνεται στις δοκιμές, τι γίνεται με τις διαδικασίες. Θα πρέπει να βρούμε πότε πρέπει να αδειοδοτούνται, πότε πρέπει να εγκρίνονται και τι γίνεται με την πρόσβαση στα στοιχεία. Διότι πρέπει να θυμόμαστε ότι όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, με τέτοιο τρόπο που να τρομάζουν οι καταναλωτές και θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα με τις κλινικές δοκιμές και τυχόν αποτελέσματα. Κυρίως αν μιλάμε για αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα σε όλους. Δηλαδή σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να γίνει, τη γίνεται τις δοκιμές στο διαδίκτυο. Αυτός ο άνθρωπος όμως ε, ίσως δεν είναι σε θέση να κρίνει σε τι συνέπειες οδηγούν τα αποτελέσματα που δημοσιοποιούνται, τι αποτελέσματα θα έχουν για την υγεία του, η υγεία της. Μόνο ένας ειδικό μπορεί να το αξιολογήσει αυτό. Ε, συνεπώς, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις κλινικές δοκιμές και όχι με τις εγκληματικές δραστηριότητες που άπτονται αυτών. Ευχαριστώ κυρία Χίμπνερ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Ρίς είναι παρόν και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Βίλμοτ για τη γνωμοδότηση που συνέταξε. Υποστηρίζει ουσιαστικά τους βασικούς στόχους της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να προωθήσουμε την κλινική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος και να έχουμε το ύψιστο δυνατό επίπεδο προστασίας των ασθενών που συμμετέχουν στις κλινικές δοκιμές. Στην έκθεσή της, η συγγήτρια μας υπενθυμίζει ότι οι κλινικές δοκιμές διενεργούνται όχι μόνο από τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά από διάφορους ερευνητές πανεπιστημιακούς και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την έρευνα θα μπορούν να διενεργούν τις κλινικές δοκιμές καλωσορίζουμε την στήριξη της εισηγήτριας για τα προτινόμενα χρονοδιαγράμματα, για την έγκριση των κλινικών δοκιμών και για τη δημιουργία εθνικών συστημάτων ταυτοποίησης, όπως ανέφερε. Το κόστος της ασφάλισης κυρίως για πανεπιστημιακή έρευνα είναι πολύ ψηλό, πολύ συχνά και δυσανάλογο σε σχέση με, τις, ε, με τα κονδύλια που διαθέτουν οι ερευνητικοί φορεί, Δεχόμαστε την πρόταση κ. να διερευνηθούν τα θέματα δεδολογικά όσον αφορά την έγκριση κλινικών δοκιμών. Υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις κατά το παρελθόν. Ποτέ δεν ήταν στόχος των προτάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξαιρούνται αυτές οι πτυχές, όπως εξήγησε ε, σαφώς και η συγγήτρια. Αναφέρομαι σε σημαντικότατα θέμα την προστασία των ανηλίκων και των ατόμων με αναπηρία, των ασθενών με κάποια αναπηρία και αδυναμία κινήσεως. Επαναλάβαμε αυτό λεξί την οδηγία, το κείμενο της οδηγίας. Δεν υπάρχει καμία μείωση προστασίας εν συγκρίση με την οδηγία. Θέλαμε να αντικατοπτήσει τη άποψη του Κοινοβουλίου που εφάνηκε από τι συζητήσει του παρελθόντο στο κείμενο. Όσον αφορά τη διαφάνεια, διαφάνεια. Συμφωνούμε την άποψη της εκθέσεως ότι χρειάζεται διαφάνεια όσον αφορά τα στοιχεία των κλινικών δοκιμών. Τίθενται διαφορετικά ζητήματα. Η διαφάνεια των κλινικών δοκιμών πρέπει να βοηθάει του ρυθμιστικούς φορείς που πρέπει να ε, δώσουν άδεια διοδότηση βάσει των στοιχείων και μετά θέλουμε διαφάνεια τα στοιχεία εν γέννη τα δεδομένα παράγονται από την έρευνα ε, και προβάλλονται τελικά και στις συνοπτικά αποτελέσματα. Για το πρώτο είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων. Υποστηρίζει πλήρως την EMA η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά τη δημοσιοποίηση τα στοιχεία των κλινικών δοκιμών που απαιτούνται για την αδειοδότηση των φαρμάκων. Για την πρόταση που συζητούμε για τη διαφάνεια εν γέννη των στοιχείων που προκύπτουν από την έρευνα έχει σημασία το τι δημοσιοποιείται ένα χρόνο μετά το τέλος των κλινικών δοκιμών. Πόσα στοιχεία θα δημοσιεύονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά την πρόταση της εισηγήτριας. Όμως όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι κανόνες που θεσπίζουμε δεν αφορά μόνο τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες αλλά και μικρά, μικρές, μικρά προγράμματα ερευνητικά πανεπιστημιακά. Οι εκθέσεις για τις κλινικές δοκιμές είναι η μορφή που τη μορφή τα στοιχεία δίνονται στην EMA ή e στους εθνικούς φορείς για την αδειοδότηση και εμπορία των φαρμάκων. Να πω κάτι για τις σπάνιες ασθένειες και τις σχετικές μελέτες. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κλινικών δοκιμών. Διότι οι συμμετέχοντες ασθενείς ε, μαζεύονται πολλά κέντρα για να γίνουν οι μελέτες. Πρέπει να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους. Βάσει του κειμένου της κυρίας Γουίλμοτ πιστεύουμε ότι θα διεξαχθούν επικοδομητικές συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία πριν τις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Ρίς. Δίνω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Γουίλμοτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα καταδαπανίσω το χρόνο που δεν έχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού που έλαβαν το λόγο και ιδίω του εισηγητέ, γιατί νομίζω ότι έχουμε μια ευρεία βάση για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Είχαμε πολλέ συναντήσει προηγουμένως προτού συγγράψω αυτή την έκθεση και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε γενικές γραμμές, όλοι θέλουμε ένα καλό νομοθέτημα. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες βέβαια και κάποιες διαφορές που μπορούμε να συζητήσουμε. Είμαι έτοιμο να συζητήσω με οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Δύο-τρία θέματα θα διεξέλθω. Οι Επιτροπέ Δημοδεοντολογία νομίζω ότι το αντιμετώπισε και το αντιμετώπισε ικανοποιητικά για όλου για το χρονοδιάγραμμα. Είναι σαφέ ότι οι περισσότερε σκιώδει υποστηρίζουν την Κομισιόν Νομίζω ότι έκανε καλή δουλειά η Κομισιόν και πρέπει να έχουμε μια πολύ στεναρή διαπραγματευτική θέση γιατί τα κράτη-μέλη θα θέλουν να παρατείνουν τις χρονικές προθεσμίες. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν ήδη χαλαρά θα καταλήξουμε με πολύ μακρά χρονοδιαγράμματα. Είναι απαραίτητο να παραμείνουμε πιστοί στην πρόταση της Κομισιόν για τα χρονικά όρια. Το θέμα της διαφάνειας. Υπήρξαν τεράστιες συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης με τους εμπλεκομένους κτλ. για τα θέματα διαφάνειας. Από τη σημερινή συζήτηση είναι φανερό ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι υπερβολικό να έχει κανείς την ε, έκθεση και μόνο. Είναι υπερβολική έκθεση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να έχουν όλα τα ακατέργαστα δεδομένα. Εγώ νομίζω ότι οι κλινικές εκθέσεις είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος τρόπος να γίνεται και θα υπάρχει φυσικά και ένα συνοπτικό σημείωμα για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να δουν όλες τις λεπτομέρειες. Είναι τεχνικό το κείμενο της έκθεσης, αλλά θα υπάρχει και ένα συνοπτικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να επαναναλυθούν και να ελεγχθούν. Πιστεύω ότι είναι μια σωστή συμβιβαστική λύση, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και ελπίζουμε ότι θα είναι φορές αυτές οι συζητήσεις, αλλά θα ήθελα να πω σε όλους του κοιόδης συζητητές, αν θέλετε να συζητήσετε κάποια πτυχή αυτού του θέματος, μιλήστε μου για να εξετάσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ευρεία συμφωνία για τα θέματα αυτά, γιατί και εγώ θέλω να ευδοκιμήσει αυτό το νομοθέτημα στην τρέχουσα νομοθετική περίοδο. Θα ήταν καλό να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία και για τους ασθενείς και για τους ερευνητές στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρο, κυρία Βουέλμποτ. Πρωτού θεσπίσουμε προθεσμία για τροπολογίε, νομίζω ο κύριο Λίζα έχει ένα διαδικαστικό θέμα. Ναι. Να ξαναπώ πω πρέπει να βάζουμε λίγο την προθεσμία για τι τροπολογίε, να το συζητήσουμε ίσω οι συντονιστέ, αλλά μία παράκληση στην κυρία Ρης. Διαβάστε το κείμενο η οδηγία του 2001, μιλάει για προστασία των παιδιών και λοιπόν ατόμων που δεν ε, έχουν ε, καταλογισμό ε, διαφορετικά από ό,τι εσείς το λέτε. Ε, είναι διαφορετική η διατύπωση της Κομισιόν και οι ειδικοί που εργάζονται πάνω σε αυτά τα θέματα μου είπαν πως νερώνει η προστασία, εξασθενεί. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο εξασθενεί και εάν θεωρεί η Κομισιόν πως είναι το ίδιο πρέπει να γράψει το ίδιο. Γι' αυτό παρακαλώ να υποστηρίξετε την τροπολογία μου που μεταφέρει αυτό το κείμενο του 2001. Κυρία Βούλμοντ, θέλετε να σχολιάσετε την πρόταση του κυρίου Λίζε. Ήδη το συζητήσαμε αυτό. Η έκθεση αυτή έχει βγει από το καλοκαίρι. Οπότε ε, πρέπει να ξέρετε τι τροπολογίες θέλετε να υποβάλλετε. Η έκθεσή μου είναι διαθέσιμη από τις 13 ε, Φεβρουαρίου και οι τροπολογίες ε, έχουν προθεσμία μέχρι τι 26. Ο καιρός επαρκεί γιατί δεν θέλω να καθυστερήσουμε τώρα, θέλω να περάσει αυτή η νομοθεσία. Ευχαρίστω να καθυστερήσει μία-δύο μέρες, αλλά θέλω να γίνει η συζήτηση των τροπολογιών στην Επιτροπή στη... την 21η Μαρτίου. Προτιμούσα να μην καθυστερήσει ένα μήνα. Κάνα δύο μέρε. εντάξει αλλά να μείνουμε εντό. προγράμματος. Αλλά ήταν ε, διαθέσιμη από τι 13 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Έχετε απολύτω δίκιο. Η πρόταση τη Κομισιόν δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2012, οπότε την είχαμε εδώ και καιρό. Τώρα, για να μείνουμε εντό χρονοδιαγράμματος για τις ε, τροπολογίες ε, και την ψηφοφορία στην Επιτροπή περιβάλλοντο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, πρέπει η προθεσμία για τις τροπολογίες να οριστεί την επόμενη εβδομάδα. Αρχικά είχε οριστεί στις 26 Φεβρουαρίου, μπορούμε να το αναβάλουμε κατά μία μέρα, αλλά αυτή είναι η μόνη καθυστέρηση που μπορούμε να επιτρέψουμε. Για να μείνουμε εντός του προγράμματος. Προτείνω λοιπόν η προθεσμία να οριστεί 27 Φεβρουαρίου τρέχοντος. και θα τα δούμε στην Επιτροπή θα τις εξετάσουμε το Μάρτιο και θα ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα τη ημερησία διάταξη ε, για την αλληλεία ε, βαθέων υδάτων και θα δώσω τον λόγο στην Άννα Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μελήσω τη μητρική μου γλώσσα. Γνωρίζω ότι πρόκειται περί γνωμοδοτήσεως για την Επιτροπή Αλίας. Δυστυχώς όμως πιθανότατα θα χρειαστεί χρειαστούν περισσότερες εξηγήσεις από την πλευρά μου, οπότε θα χωρίσω την παρέμβασή μου σε τρία τμήματα. Πρώτα απ' όλα θα ενημερώσω σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα ήθελα να πω κάτι περί της αλίας σε βαθαία ύδατα και ποιες είναι οι συνέπειες και μετά να αναφερθώ γενικά στην όλη γνωμοδότηση. Όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο υφιστάμενος κανονισμός για την αλληλεία στα βαθαία υδάτα, κυρίως στον Ατλαντικό, στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, είναι κάτι που ισχύει για την τελευταία δεκαετία. Η νομοθεσία στον τομέα αυτό δεν κατέστησε δυνατό να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες για την αλληλεία και το βανθυπελαγικό περιβάλλον και το, την βανθυπελαγική πανίδα αυτά τα χρόνια. η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλό, καλή προσπάθεια να ληφθεί υπόψη η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοπικιλότητας στα πλαίσια της διαχείρισης ε, της αλίας υδάτων. Η επικοινότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλουμε να έχουμε βιώσιμη αλία των βενθοπελαγικών ειδών και να μειώσουμε και τον αντίκτυπο της αλίας βαθέων υδάτων στα βενθοπελαγικά αυτά είδη. Θέλουμε να αυξήσουμε και την επιστημονική μας γνώση όσον αφορά τα μεθοπαλλαγικά είδη και πώς ζουν. Αυτά για την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω τώρα τι είναι η αλία βαθέων υδάτων. Τα βενθοπελαγικά είδη και και το οικοσύστημα των βαθέων υδάτων είναι από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς και οι ερευνητές έχουν εκθέσει, έχουν ερευνήσει μόνο μικρό ποσοστό του τομέα αυτού. Υπάρχουν χιλιάδες είδη για τα οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα. Στα 4.000 μέτρα, σε τέτοιο μεγάλο βάθος, σε αυτό το περιβάλλον ε, υπάρχουν πολλά γνωστά είδη. Και κοράλια. Μερικά από τα κοράλια μπορεί να έχουν και ηλικία μέχρι και 8.000 έτη. Ε, ε, και λόγω της πίεσης και της θερμοκρασίας σε αυτά τα βάθη τα είδη είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Αναπαράγονται αργά στη ζωή τους, μπορούν να ζήσουν και μέχρι ηλικία 150 ετών εκτίθεται πολύ στην υπεραλία και πολλά είδη έχουν υπεραληφθεί. Ο τόνος και ο βακαλάος που είναι κοντά στις ακτές ε, έχουν υπεραλειφθεί και οι ψαράδες βγαίνουν πιο ανοιχτά, πάνε σε μεγαλύτερο βάθος για να βρουν ψάρι. Ε, οι αλείς έχουν ειδικό εξοπλισμό για να μπορούν να ψαρεύουν κάποια είδη και μπορούν να φτάσουν καμιά φορά μέχρι σε βάθος 2 ε, χιλιόμετρων. Η αλία για τα βενθοπελαγικά είδη οδηγεί σε ανεπανόρθωτη ζημία στο περιβάλλον το βενθοπελαγικό και χάνονται και κοράλια και οι τράτες που αλλιεύουν σε βαθύ είδωρ ε, κάνουν μεγάλη ζημιά γιατί σέρνεται το δίχτυ η τράτα στο, στο βυθό, παρασύρει τα πάντα και μετά μέχρι 30% των αλλιευμάτων απορρίπτονται διότι δεν έχουν εμπορική αξία και κανένα από τα απορρίμματα, από τα είδη που απορρίπτονται δεν μπορεί να επιβιώσει γιατί απορρίπτονται σε βάθος λανθασμένο. Αυτά λοιπόν για αυτού του είδους την αλία. Τι μπορούμε να κάνουμε μετά, αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της παρέμβασής μου. Τι μπορούμε να κάνουμε μέσω του κειμένου και μέσω της εκθέσεως. Υποστηρίζω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πράγματι τονίζω ότι υπάρχει ανάγκη για πιο συνετή προσέγγιση όσον αφορά τη θέσπιση νομοθεσίας για την αλία βαθέων υδάτων μεγάλου βάθους ε, για να προστατεύσουμε τα πολύ ευάλωτα ε, είδη και το οικοσύστημα. Προτείνω λοιπόν να έχουμε καλό ορισμό των ευαλώτων θαλασσίων οικοσυστημάτων θα πρέπει να συμβάλλουμε στο να σταματήσει η απώλεια της βιοπικιλότητας, κάτι που διαπιστώνεται τώρα. Προτείνω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει την πρότασή της για να ευθυγραμμιστεί με τη συνθήκη της Αβώνας, όπου λέει ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να εντάσσεται στη σύνταξη, θέσπιση και εφαρμογή νομοθεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να πετύχουμε ε, βιώσιμη αλία. Εγώ θα αναφερόμουν και σε διεθνείς συμφωνίες σχετικές. Έχουμε και το ψήφισμα της συνέλε, ε, του, των Εθνών για την ε, αλία σε βαθέα ύδατα και την προστασία των ειδών. Υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιοριστεί η ζημία που προκαλούμε μέσω εξοπλισμού που προξερεί βλάβες θα πρέπει να αλλάξει ο εξοπλισμός εντός ενός έτους και θα πρέπει να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε αλία μεγάλου βάθους για τα λευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που κινούνται εντός των υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού διότι είναι μια παγκόσμια εμβελίας δραστηριότητα και χρειάζεται και συντονισμός μας με τις τρίτες χώρες ε, τρίτες χώρες που ασχολούνται με την αλία μεγάλου βάθους και θα πρέπει να θυγραμιστούμε και με τις ανάλογες διεθνείς συμφωνίες. Θέλω να υποβάλω τροπολογία για την αλία τρίτων χωρών σε βα... βαθαία ύδατα. Προτείνω να δούμε και ποιες είναι οι συνέπειες της αλίας σε μεγάλο βάθος. Ε, σύμφωνα με τις ιδέες του ΟΗΕ, προτείνω επίσης να δούμε και ποιος είναι ο αντίκτυπος της αλίας για τους υφιστάμενους αλληλευτικούς χώρους και όχι τα νέες περιοχές. Λοιπόν, έχουμε τρία σημεία να εξετάσουμε σε 7 λεπτά, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο μόνο στους δύο παρόντες κοιόδης για ένα λεπτό για αυτό το θέμα. Είδε ΔΕΜΗ δεν έχουμε δυνατότητα να εξαντλήσουμε τη μέσα διάταξη. Λίντα, λοιπόν, έχει το λόγο. Απλώς να πω ότι υποστηρίζω την Άννα Ρόσπαχ στην πρότασή τη. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία για τα θέματα αυτά. Πριν από δύο εβδομάδες ψηφίσαμε υπέρ της προστασίας των αλλιευμάτων για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε την πολιτική σε μεγάλο βάθος χωριστά και αυτό υποστηρίζω την ΑΡΟΣΠΑ Κυρία Κοκοβίτσου. Χωρίς μικρόφωνο. δεν θέλει να λάβει το λόγο. 22 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε 20 και 21 Μαρτίου και αν θέλει ο Θεός τον Απρίλιο στην Επιτροπή Αλίας και τον Ιούνιο στην Ορομέλεια. Επόμενο θέμα, πάλι αναρόσπαχ για την ε, περιφερειακή στρατηγική για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ όμως αυτή τη φορά να είστε πιο σύντομοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα υπερβολικά σύντομη αυτή τη φορά. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω, στο οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι. Πρόκειται λοιπόν εδώ πέρα για μια νομοδότηση που απευθύνεται στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά τη βιομηχανι... τις βιομηχανικές ζώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προτείνω λοιπόν αν ε, βάλουμε κάποια περιβαλλοντικά ζητήματα στρατηγική αυτή όπως ε, τον καθαρισμό ε, μολυσμένων περιοχών και υδάτων. Είναι λοιπόν μια ολοκληρωμένη περιοχή Θα προτείνω κάποιες προσθήκες και ελπίζω και οι συνάδελφοι να συνεισφέρουν με επικοδομητική κριτική. Εγώ κατάγομαι από μια χώρα όπου είναι κάτι το φυσιολογικό να μην είναι στη μέση κατοικημένων περιοχών οι δημοφανικές περιοχές. Και εσείς το ίδιο κύριε Πρόεδρε, αλλά υπάρχουν χώρες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ο κόσμος ζει πάνω από το εργοστάσιο. Το είδαμε αυτό όταν είδαμε και την ε, οδηγία σε Βέζο. Πρέπει λοιπόν να γίνουν πολλά ακόμα. Και αυτό θεωρώ πως είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία είναι μη νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας. Αν κάποιο άλλο σκιώδης ε, θέλει να πει κάτι, σύντομα θα δώσω το λόγο. Κύριε Χιμπνερ, ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι καλό που ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση όσον αφορά την περιφερειακή στρατηγική για τι βιομηχανικέ περιοχέ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια τίθενται κάποιε προτεραιότητε. Πρώτα απ' όλα η χρηματοδότηση. Και εδώ μπορούμε να μιλάμε για συγχρηματοδότηση και από τα κράτη και ε, από, σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο και διαθροτικές αλλαγές αυτού αυτούς τους Και υποστηρίζουμε την τοπική μικρή βιομηχανία που θα μπορούσε να γίνει πιο καινοτόμα και πιο καθαρή. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ε, στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των περιφερειών, αλλά μπορεί να διαφέρουν τόσο πολύ που είναι ανέφικτο να χρησιμοποιηθεί η ίδια τεχνολογία. Θα πρέπει λοιπόν καταρχάς να εστιαστούμε επί, νέων καθαρών τεχνολογιών και να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές όταν αυτό είναι οικονομικά βιώσιμο και εφικτό. Βεβαίως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεγαλύτερο μερίδιο να κατέχουν και αυτό χρειάζεται να γίνει και θα πρέπει να υπάρξει και συμμόρφωση με σχετικού κανονισμού. Έχουμε κανονισμού όσον αφορά την καθαρότητα των υδάτων, τα απόβλητα κλπ. Άρα θα πρέπει να δούμε και αυτό εδώ που είναι σημαντικό. Ε, επόμενο, η καινοτομία ε, όσον αφορά την αποθήκευση ε, των ανασύμων πηγών ενέργειας. Γιατί για την ώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε σωστές μεθόδους για την αποθήκευση ανανοσίμων πηγών ενέργειας, δεν έχουμε κίνητρα επίσης για ε, καινοτομίε στον οικολογικό τομέα, μετά ολοκληρωμένες μεταφορές. Θα πρέπει να έχω στη διάθεσή μου λίγο χρόνο παραπάνω. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα των μεταφορών, είναι σημαντικότατο. Και τέλος, το σημαντικότερο, με τη συμμετοχή των πολιτών μπορούμε να δημιουργήσουμε περιφερειακή πολιτική ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν κάποια καθήκοντα, αλλά να έχουν και πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων περιφερειακών και σε άλλα επίπεδα. Είναι σημαντικό λοιπόν οι πολίτες να μπορέσουν να συμμετέχουν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που καταφέρατε να... Ευχαριστώ στους διερμηνείς που ακολούθησαν σε αυτή την ταχύτητα, λέει πρόεδρος. Λίντα, να πω κάτι κι εγώ, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι υποστηρίζω και πάλι αυτά που μας συνέγραψε η Αν Χόσπακ για την ε, ενεργειακή απόδοση, πόσο σημαντική είναι αυτή για να καταπολεμηθεί η ανεργία σε βιομηχανικές περιοχές, μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας επενδύοντας σε αποδοτική χρήση της ενέργειας και να βοηθήσουμε και τον κόσμο να κάνει οικονομίες. Δεύτερον, κάτι που δεν αναφέρεται και αφορά το ρόλο των κρατικών ενισχύσεων για να βοηθηθούν οι, βιομηχανικές ε, περιοχέ δημιουργήσεω τη απασχόληση και επενδύσει. Στην Επιτροπή Ενεργική Πολιτική συζητήσαν ένα νέο ε, ένα κατευθυντήριε γραμμέ για αυτή την πολιτική. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν επιτρέπεται σε βιομηχανικέ περιοχέ να δώσουν κρατική ενίσχυση σε μεγάλε εταιρείε. Είναι λάθο, γιατί κάποιε μεγάλε εταιρείε μπορούν να ερευνήσουν ε, νέε τεχνολογίε και αποδοτικέ χρήσει ενέργεια να δημιουργήσουν απασχόληση, θα το ξανασκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ θα υποβάλω σχετική τροπολογία. Και εσεί, κύριε Παναγιώτοφη, σχεδόν για του φιλελευθέρου και συγκητή για, για το νέο θέμα. Έχετε λεπτά. Τι θέλετε να χρησιμοποιήσετε εδώ ή στο άλλο θέμα για την έκθεση για, ε, του ισορρευτέ. Αμέσω για την έκθεση αυτή, λοιπόν, για του ισορρευτέ. Θα είμαι. Πάρα πολύ σύντομο. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλους τους σκιώδησίητες, όλους που με υποστήριξαν και έχουν καταθέσει μια σωρία τροπολογιών. Δεν θα μακρηγορήσω. Δύο λόγια μονάχα. Έχω προτείνει ότι η άρση της εξαίρεσης να καθυστερήσει για ένα χρόνο και να φτάσει στο τέλος του 2016. Έχω εξηγήσει στην Επιτροπή μας γιατί το ζητώ αυτό. Εγώ προσλέπω στις ε, συζητήσεις με τους κοιόδης συζητητές πριν από την ψηφοφορία το Μάρτιο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λογική συμβαστική θέση μεταξύ των διαφόρων απόψεων για να προστατεύσουμε και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε όλη την αλυσίδα προσθέμενης αξίας ενώ συγχρόνως εξασφαλίζουμε την προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και δίνοντας τη δυνατότητα να υπάρξει τεχνολογική ε, ανάπτυξη, διαμοιρασμός βελτίστων πρακτικών κτλ. στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ η προθεσμία τροπολογιών 26 του μηνός, 20 Μαρτίου ψηφοφορία. Κυρία Κούκορη, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, με σκιώδης για αυτή την έκθεση. Δεν έχουμε αρχίσει με τις μπαταρίες ακόμα. Α, ναι, με τις μπαταρίες. Απασχολούμαστε τώρα. 26 Φεβρουαρίου και 20 Μαρτίου για, τους, για τις βιομηχανικές περιοχές και μετά είμαστε στις μπαταρίες. Έχετε τον λόγο. Τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους μου από το ΕΛΚ. Ε, εγώ άκουσα τα ειδικά. Τώρα για τις μπαταρίες τελικά θα μιλήσετε. Εγώ νόμιζα θα μιλήσω για τις μηχανικές ζώνες. Δύο λόγια. Ε, το θέμα αυτό. Πρέπει να βρούμε την καλύτερη λύση για να εξορροπήσουμε βέβαια σε επιδράσεις στο περιβάλλον και στην υγεία με ε, τις επιδράσεις στη βιομηχανία λόγω της αλλαγής της οδηγίας. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε πως ε, είμαστε ακόμα σε καιρό κρίσης. Ε, η κρίση είναι ακόμα εδώ. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ κάποιων τροπολογιών που είναι, δεν είναι πολύ ρεαλιστικές. Ελπίζω τις ε, μπαταρίες με υδράργυρο να, ε, να μην εκτίθενται τα παιδιά σε αυτές. Και ελπίζω σιγά σιγά να αναφερθούν και αυτές και οι μπαταρίες νικελίου καδμίου. Για τη συλλογή τώρα και την ανακύκλωση ε, πρέπει να το δούμε ως ένα πόρο. Γιατί Είμαι σίγουρη πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο αυτές οι πρώτες Ευχαριστώ. The next Dan is not here. Dan δεν είναι εδώ. Τον αντικαθιστάτε εσείς. Λίντα. Ναι, να πω πως η ομάδα μας δεν συμφωνεί με την επέκταση των προθεσμιών. Δεν υποστηρίξαμε την επέκταση για τα ηλεκτρικά εργαλεία ούτε και τώρα. Ούτε την προηγούμενη φορά ούτε και τώρα. Ε, καλωσορίζουμε μετά του Διενεργύρου, αλλά ο κύριο Γιώργενσεν θα καταθέσει τροπολογίε. Εγώ όμω και για του πράσινου, λέει ο πρόεδρο, και εγώ θέλω πιο σύντομε προθεσμίε ε, για τον Υδράργυρο. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Η εξαίρεση αυτών των εργαλείων δεν χρειαζόταν ούτε την προηγούμενη φορά, ούτε τώρα χρειάζεται. Δεν είναι πλέον αναγκαία. Και επίση για το πόσο εύκολα μπορούν να αφαιρεθούν, γιατί Κοιτάξτε, μειώνεται ο χρόνος ζωής ε, γιατί έχει καταστραφεί η μπαταρία. Όχι, πρέπει οι καταναλωτές να μπορούν να αλλάζουν την μπαταρία ακόμα και αν είναι ενσωματωμένοι για να μην ε, κοντένει ο κύκλος ζωής από μια βλάβη της μπαταρίας. Αυτά οι υπόλοιποι ισχυώδεις λείπουν, οπότε μπορούμε να τελειώσουμε αυτή τη συνεδρίαση με 5 λεπτά καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνεδρίαση, θα, η ψηφοφορία μου συγχωρείτε, θα είναι στις 20 Μαρτίου. Ευχαριστώ. So we will continue at 3 o'clock with the hearing uh, for the candidate for the director of EEA. See you.